Good afternoon, colleagues. I don't think I need to use the hammer to begin the <laughs> meeting today. Um, so following on our important votes on... Uh... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα... να σας πω ότι σήμερα το πρωί είχαμε ξεκινήσει τις εργασίες warmly welcome the director of the EMC. Και συνεχίζουμε λοιπόν τώρα με την υποκειμενική μας συνεδρίαση και σε αυτήν την ε, συνεδρίαση έχουμε καλέσει τον, τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Ταξικομανίας για έτσι ώστε να μας προσθέσει τη διάσμη του 2017 σχετικά με την έκθεση για τα ναρκωτικά Περιλαμβανομένη έκθεσης τάση και εξελίξει του αστικού δελτίου για το 2017 και των 30 εκθέσεων χωρών σχετικά με τα ε, ναρκωτικά. Σας έχουν ήδη δοθεί ε, αντίγραφα της έκθεσης και επομένως θα δώσω αμέσως τον ε, λόγο στον καλεσμένο μας για μια σύντομη παρουσίαση και μετά βεβαίως θα δώσω το λόγο στα πολυπληθή μέλη τα οποία έχουν κατακλείσει την αίθουσα. Λοιπόν, να συνε... εντάξει, ελπίζω ότι θα έρθουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι μετά. Ο μιλητής μας θα μιλήσει για 10 ε, λεπτά. Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μεγάλη χαρά ε, που βρίσκομαι σήμερα εδώ έτσι ώστε να σας παρουσιάσω τις κεντρικές γραμμές ε, της έκθεσης. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, υπάρχει μια πολύ σημαντική δέσμη ε, πληροφοριών η οποία συνοδεύει την έκθεση γιατί εμείς παρουσιάζουμε μαζί με την έκθεση και ένα αναλυτικό στατιστικό δελτίο όλων των των ε, στατιστικών. Και επίσης, πρώτη φορά φέτος, έχουμε και ένα νέο μορφότυπο που αφορά εκθέσεις αναχώρα έτσι ώστε να έχουμε και μία συνολική έποψη των καταστάσεων, ε, ε, των εθνικών καταστάσεων. Και να πω ότι κάθε έκθεση παρουσιάζει και ένα τμήμα όπου εντάσσει την κάθε μία χώρα στο γενικότερο ε, πλαίσιο. Ε, είχαμε κάποια πρώτα κεντρικά ε, στοιχεία τα οποία έχουμε παρουσιάσει. Ενδεχομένως θα ξέρετε ε, ότι το MCDD είναι επικεφαλής φέτος του δικτύου για τα ναρκωτικά και θα ήθελα και εξ και των Γενικών Διευθύνσεων Ασφάλεια και δικαιοσύνη θα ήθελα να εκφράσω τον αποτοπιασμό μου για, ε, για τα, τα πρόσφατα τρομοκρατικά ε, χτυπήματα. Ποια είναι τα κεντρικά στοιχεία της νέας έκθεσης. Ε, εγώ θα ασχοληθώ με πέντε κεντρικά στοιχεία και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. Τα πέντε οι πέντε μεγάλες ε, αλλαγές ε, έχουν να κάνουν με την αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση, overdose. Επίσης, ε, αυξανόμενη απειλή για την υγεία. Τρίτο στοιχείο κεντρικό είναι ότι υπάρχει ένα ζήτημα, είναι ένα ζήτημα το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, νέες ουσίες, Μιλάμε για νέες ψυχοτρόπες ε, ε, ουσίες και είναι σημαντικό που σήμερα το πρωί ε, υπήρξε αυτή η σημαντική ψηφοφορία που θα μας δώσει τη δυνατότητα να μελετήσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό. Πέμπτο στοιχείο είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια διαπιστώσαμε αύξηση στη διαθεσιμότητα της κοκαίνης. Τελευταίο δε σημείο το οποίο θα θίξω ε, ε, ή θα αφορά κάποια νέα στελέχη της ε, κάνοβης. Χρήση και κατάχρηση των στελεχών αυτών. Να ξεκινήσω με τους θανάσους τους από υπερβολική δόση, overdose, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά βλέπουμε ότι υπάρχει αυξανόμενο ποσοστό θανάτων σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά. Αυτό που είναι σημαντικό και νομίζω είναι σημαντικό και για εσάς ως μέλη της Επιτροπής σας εδώ είναι ότι η περισσότεροι από τους θανάτους αυτούς σχετίζονται με οπιοειδή και με ηρωίνη, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις όμως ε, συνδυάζονται και με άλλες ουσίες. Αυτό που μπορείτε να παρατηρήσετε και θα το δείτε και σε αυτές τις διαφάνειες που βλέπετε, ε, οι πράσινες στήλες είναι ότι παρά το γεγονός ότι ε, διαπιστώνουμε ότι τα οπιοειδή και οι ηρωίνη χρησιμοποιείται περισσότερο, ε, ε, αυτό που μας, ε, το νέο στοιχείο είναι ότι οι χρήστες ανήκουν όλο και σε πιο μεγάλες ηλικιακέ ομάδες σε σχέση κυρίως με το 14 και το 2015. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι τα τελευταία χρόνια είδαμε στην Ευρώπη και στο γενικότερο ευρωπαϊκό χώρο Διαπιστώνουμε λοιπόν αύξηση των υπερβολικών θανάτων από υπερβολική δόση ε, και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Δύο ειδών είναι οι παρεμβάσεις. Πρώτον, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε τέτοιες ε, overdose ε, και δεύτερον να βρούμε τον τρόπο σε περίπτωση υπερβολικής δόσης να επιβιώσει το, το άτομο. Ε, και ε, υπάρχουν ήδη κάποια εναλλακτικά, ε, κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι με βάση τις θεραπείες με οποίο ήδη υπάρχουν τέτοια σχετικά προγράμματα στην Ευρώπη. Δεύτερο στοιχείο το οποίο αυξάνεται είναι τα νέα συνθετικά οποίο ήδη και η σημασία προγραμμάτων αναλοξών που έχουν την, δίνουν την δυνατότητα ε, στα άτομα να ξεπεράσουν την υπερβολική δόση. Και ε, σε 7 χώρες ε, υπάρχει η λύση των δωματίων κατανάλωσης ναρκωτικών ελεγχόμενων, drug consumption rooms. Υπάρχουν 78 λοιπόν τέτοιου είδους θηρίδες και ξέρουμε ότι παρόμοιες λύσεις ε, υπάρχουν και σε άλλες χώρες εκτός Ευρώπης, στον Καναδά ας πούμε έτσι ώστε να ξεπεραστεί η νέα επιδημία της χρήσης των οπιοειδών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως να χρησιμοποιηθεί εναλλακτική ε, ε, μορφή αυτών των εναλλακτικές ιατρικές θεραπείες όπως η μεθαδόνη και άλλες και όλο αυτό όλα αυτά τα στοιχεία αφορούν τη συνολική δέσμη του προβλήματος. Δεύτερον, δεύτερο πρόβλημα είναι τα νέα συνθετικά οπιοειδή πρόκειται για μια αυξανόμενη απειλή υγείας. 25 νέα τέτοια ε, είδη συνθετικών οπιοειδών έχουμε ταυτοποιήσει ε, τα τελευταία χρόνια. Ε, πέρσι δε μονάχα 8 ε, επίσης βλέπουμε ότι και σε άλλα προϊόντα υπάρχει υψηλή συγκέντρωση τέτοιων προϊόντων, ε, πράγμα που σημαίνει ότι ε, λόγω τυχαίας έκθεσης μπορεί να προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Οι φεταμίνες επίσης ε, είναι ένα πρόβλημα τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για μια οικογένεια φαρμάκων πάρα, ουσιών πάρα πολύ ισχυρών. Ε, κυρίως χρησιμοποιούνται για αναισθησία και έχουν και αναλγητική δράση αλλά ε, έχουν, έχουμε πάρα πολλές ε, παρατηρήσεις τέτοιου για τέτοια προϊόντα στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης. Οι ουσίες αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές γιατί όπως είπα και προηγουμένως έχουν βρεθεί τα τελευταία δύο-τρία χρόνια όχι μονάχα ε, ε, στην καθαρή τους φαρμακευτική μορφή αλλά ε, και σε αναμίξεις με κοκαίνη και ηρωμίνη πράγμα που σημαίνει ότι αυξάνεται πολύ ο τίνος υπερβολικής δόσης. Σημαντικότερος λοιπόν, υψηλότερος ο κίνδυνος και βλέπουμε ότι και στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες πολλοί άνθρωποι του star system, μουσική κλπ. Ε, έχουν χρησιμοποιήσει ε, τέτοιου είδους ε, ουσίες χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι τις καταναλώνουν. Ε, αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι και 300 φορές πιο ε, δυνατές από την μορφήνη. Τρίτο έβριμα αφορά ε, την χρήση νέων και την εξέλιξη νέων ψυχοτρόπων ουσιών. Ε, υπάρχει μία μείωση της ανιχνεύσης, αλλά η διαθεσιμότητα εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ ε, υψηλή. Να σας πω, το 2016 ε, είχαμε ανιχνεύσει 66 νέες ουσίες. Έχουμε λοιπόν μία μείωση σε σχέση με την κορυφή που είχαμε πιάσει το 2014. Ε, θα πρέπει να δούμε βεβαίως και ποια θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, της ε, νέας νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα, γιατί διαπιστώνουμε ότι και στην Κίνα υπάρχει τροποποίηση των κανόνων και επομένως πρέπει να περιμένουμε να δούμε. Ωστόσο, έστω και αν ο αριθμός των ανιχνευθέν ανιχνευτισών συγγνώμη, ουσιών ε, έχει ε, μειωθεί. Υπάρχουν ε, στην αγορά ουσίες οι οποίες είναι πολύ πιο δυνατές και πολύ πιο επικίνδυνες. Αν δει κανείς δε το σύνολο του, ε, ε, του καλυπτόμενου το EMCDDA ε, περιβάλλον είχαμε 423 ουσίες οι οποίες είχαν ανοιχνευτεί μόνο το 2016. Το ζήτημα δηλαδή δεν είναι μόνο να ξέρουμε ποιες είναι οι νέες ουσίες αλλά και ποια είναι η εξέλιξη των παλαιών ουσιών και πόσο μεγαλώνει η διαθεσιμότητα ουσιών στην αγορά. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι, και αυτό από μόνο του καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η απόφαση που πήρατε σήμερα το πρωί. Υπάρχει και ένα νέο φαινόμενο και υπάρχει και μία σύντομη δημοσίευση ε, σχετικά με την χρήση υψηλού κινδύνου σε περιθωριοποιημένους ε, πληθυσμούς ε, και εδώ βλέπουμε ότι ε, έχουμε πολύ συχνά ε, τους χρήστες οπιοειδών την έγχυση ε, κατηνοειδών που είναι ένα που είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπουμε πολύ συχνά, ε, κυρίως σε άστεγους. Οι άστεγοι χρησιμοποιούν επίσης πολύ συχνά και συνθετικά ε, ε, προϊόντα κάναβης. Και επίσης και στις φυλακές έχουμε δει ότι τέτοιου είδους χρήστες αυξάνουν. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια έχουμε διαπιστώσει και αύξηση της ε, χρήσης ε, κοκαίνης. Ε, έχουμε πολλές, πολλούς δείκτες οι οποίοι συνδύνουν στο συμπέρασμα ότι είναι πιο εύκολα διαθέσιμη η κοκαίνη και επίσης ότι είναι και πιο καθαρή η μορφή της κοκαίνης η οποία βρίσκεται διατίθεται στην αγορά. Γι' αυτό και φέτος και στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε να παρατηρήσουμε εάν αυτή η αυξημένη διαθεσιμότητα ε, τελικά ε, ε, οδηγεί και σε περισσότερους θανάτους. Θα δούμε, το βλέπουμε και στις αναχώρα εκθέσεις ότι υπάρχουν συγκεκριμένες χώρες και μάλιστα συγκεκριμένες πόλεις οι οποίες πρέπει να παρακολουθηθούν με μεγαλύτερη προσοχή. βλέπουμε ότι υπάρχουν ότι, ότι τις 33 χώρες οι οποίες ε, συμμετέχουν στην ανάλυση των, αποβλ, των υγρών αποβλήτων ε, που έχουμε κάνει, ε, στις 33 αυτές χώρες έχουν αυξηθεί τα κατάλοιπα της κοκαίνης. Η κάναβης τώρα είναι το ναρκωτικό το οποίο έχουν χρησιμοποιήσει, του έχουν πάρει τουλάχιστον ε, τα μεγαλύτερα ποσοστά ενηλίκων ε, χρηστών ε, στην Ευρώπη τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. 87 και παραπάνω εκατομμύρια Ευρωπαίοι ενήλικες έχουν τουλάχιστον μία φορά δοκιμάσει κάνοβι και 1% των ε, ε, ε, ενηλίκων κάνουν καθημερινή χρήση. Προσπαθούμε τώρα να δούμε και τις διαφοροποιήσεις αναχώρα, καθώς επίσης και ποιες είναι οι συγκεκριμένες πληροφορίες τις οποίες μπορεί να βρει κανείς όσον αφορά την κάναβη. Πάντα σε σχέση με την κάναβη, αυτό που έχουμε παρατηρήσει είναι ότι ότι η χρήση κάναβης ε, μεταξύ φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι στο 50% της αντίστοιχης χρήσης φοιτητών ε, στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ωστόσο, η κατανάλωση αλκοόλ είναι δύο φορές μεγαλύτερη στην Ευρώπη και φτάνει στις τέσσερις φορές μεγαλύτερη κατανάλωση όταν μιλάμε για προϊόντα καπνού. Ε, υπάρχουν ε, βέβαια και ε, αυτό που προσπαθώ να καταλάβουμε τώρα είναι ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αυτές τις καταναλώσεις και γιατί είναι τόσο ισχυρή και ανθεκτική η χρήση της κάναβης. Σε γενικέ γραμμέ μπορώ να σα πω και συμπεράσματι ότι η κατάσταση όσον αφορά τα ναρκωτικά ε, είναι εξαιρετικά δυναμική και εξελίσσεται. Και επομένω ε, είναι πάρα πολλέ ε, οι αλλαγέ και οι οποίε λαμβάνουν χώρα με ταχύ ρυθμό. Επίσης, τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη έχουμε πολύ, σημαντικές, πολύ σημαντικά αποτελέσματα ε, όσον αφορά την ανταπόκριση των ε, συστημάτων ε, υγείας, των δημοσίων συστημάτων υγείας. Έχουμε επίσης και κοινά στοιχεία, διασταυρούμενα μάλλον, με τα στοιχεία για την υπατήτητα γάμα κλπ. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει επίσης είναι και η εξέλιξη της αγοράς όσον αφορά τις ψυχοτρόπες ουσίες. Αναφέρθηκα σε αυτό στην αρχή της παρέμβασής μου. Έχουμε επίσης ε, και την ε, παρουσία νέων ε, χριστών και στις έρευνες γενικού πληθυσμού βλέπουμε ότι 4 με 6% των νέων δηλώνουν ότι έστω περιστασιακά κάνουν χρήση αυτών των ουσιών. Έχουμε επίσης ε, τις τεχνικές, ε, τα, τεχνητά οπιοειδή που έχουν κατακλείσει πλέον την αγορά. Νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση απαιτεί ε, μεγαλύτερη συνεργασία και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ο Επίτροπος έχει ανακοινώσει μάλιστα και ένα νέο σχέδιο δράσης και αυτό θα αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Μπορεί μάλιστα και πριν το τέλος της ε, τωρινής Προεδρίας ε, να γίνει η ανακοίνωση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλή συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη ο τρόπος με τον οποίο εμείς ε, ε, συμβάλλουμε ε, στην όλη διαδικασία είναι μέσω της καλύτερης πληροφορήσης. Της καλύτερης πληροφόρησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και έχω χαίρομαι που είχατε πιο πολύ χρόνο από την προηγούμενη φορά για να τα παρουσιάσετε αυτά. την τελευταία φορά είχαμε πολύ έντονη χρονική πίεση και ήταν πιο εκτενή η σημερινή παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. να δώσω το λόγο στα μέλη. Στον κύριο Μπόνη, καταρχάς, που είναι ο εισηγητής μας. Thank you very much. Ε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την ε, καλή αυτή παρουσίαση και την περιγραφή κάποιων τάσεων που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τις έχουμε υπόψη και να τις κατανοούμε. Είναι σημαντικό να έχουμε υπόψη μας όλα τα φαινόμενα σε σχέση με τα ναρκωτικά και σε σχέση με τις εξελίξεις τη χρήση των ναρκωτικών στην Ευρώπη. Και ασφαλώς θα παρουσιάσω και κάποιες ανησυχίε που έχω. Καταρχάς, ότι αφορά τον αριθμό των θανάτων. Είναι δυστυχώς αυτής η και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι καλύτερες οι αντιδράσεις κυρίως ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη για την ε, γνωστοποίηση και την προώθηση του μηνύματος του πόσο επικίνδυνα είναι τα ναρκωτικά. Σημαντικό είναι να έχουμε υπόψη μας και κάποια καινούργια φαινόμενα και να λαμβάνουμε υπόψη πώς ε, μπορούμε σε κοινωνικό επίπεδο να περάσουμε σε κάποια ζητήματα. Αναφερθήκατε στις φυλακές, στους ε, φυλακισμένους, ε, στους άστεγους μιλάμε για μια νέα γενιά όταν αναλύουμε τη χρήση της κάναβης. Υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις και κάποια πρόοδο στις ΕΠΑ, αλλά Αυξάνεται η χρήση κάναβης ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προωθήσουμε λοιπόν πληροφορίες και σαφή μηνύματα από, το, από την ε, δημόσια σφαίρα για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα άτομα και να προστατεύσουμε από νέους τύπους ναρκωτικών. Κατά δεύτερον, αναφερθήκατε στην όλο και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κοκαίνη. Θα πρέπει, θεωρώ, να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την ε, προώθηση, αλλά και την πιο δυναμική παρέμβαση των σώματων της αστυνομίας, του δικαστικού σώματος κτλ. στην Ευρώπη. Γιατί τίφεται το θέμα της χρήσης, αλλά και της διαθεσιμότητας ε, των ε, ναρκωτικών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν ε, οργανώσεις, εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες και παρά διαθέτουν στην εμπορία τα αρκωτικά αυτά. Με απλό τρόπο κατά πάσα πιθανότητα. Και θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν το μήνυμα ότι μπορούμε να αντιδράσουμε. Όταν μιλάμε για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες, Ασφαλώς, όπως είπατε. Η διαθεσιμότητα εξακολουθεί να είναι υψηλή, αλλά ενδεχομένω ο αντίκτυπος ε, να είναι χαμηλότερο σε σχέση με πριν από κάποια χρόνια το 2014 που ήταν ε, στο Zenith. Αλλά είχαμε το 2016 66 νέες τέτοιες ουσίες. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να εφαρμοστούν ε, με ταχύτητα αυτές οι προτάσεις. Το μοντέλο που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την Επιτροπή και το Συμβούλιο μετά από δύο-τρία χρόνια σε αδιέξοδο που περάσαμε. Προσπάθησα λοιπόν ε, να καταμετρήσω και να αξιολογήσω τους παράγοντες αποτελεσματικότητας. Την προηγούμενη φορά καταφέραμε σε 84-85 μήνες να πετύχουμε αποτελέσματα. Τώρα μιλάμε για 36-38 μήνες. για την γρήγορη δηλαδή εφαρμογή των μέτρων για κάποιες ουσίες. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. χρειάζεται λοιπόν για να ξεκινήσετε με τον νέο κανονισμό. Υπάρχουν κάποιε προδιαγραφέ και απαιτήσει σε ό,τι αφορά τι υπηρεσίε για την κατάρτιση τη αρχική έκθεση και τη αξιολόγηση ε, κινδύνου. Και νομίζω επίσης ότι ένα από τα πλέον εκτίματα των αυτών λύσεων είναι αν δοθούν τα σχετικά μηνύματα και προτιμάσει σχετικό νομοθέτημα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η απαγόρευση των ουσιών θα είναι για όλα τα κράτη-μέλη, όχι μόνο για κάποια εξ αυτών. Και μιλάμε και για ψηφιακές οδούς. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε από αυτή την άποψη. Το τελευταίο θέμα έχει να κάνει με το μέλλον. και με τη στρατηγική σας για το 2025, τη μελλοντική στρατηγική. Γιατί αν ξεκινήσουμε τις εργασίες για τον προϋπολογισμό μετά το 2020, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστή πηγή χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της, ε, του, της υπηρεσίας. Πώς θα προθεθούν λοιπόν καλύτερα τα πράγματα, πώς θα καταπολεμήσουμε κάποια νέα φαινόμενα όπως είναι η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα παροχής ε, και εμπορίας κοκαίνης μαζί με την Europol. Τι χρειάζεται για να εφαρμόσουμε καλύτερους ε, κανονισμούς πλαίσιο για την καταπολέμηση των νέων ψυχοτρόπων ουσιών και μελλοντική στρατηγική και μελλοντική ικανότητα των υπηρεσιών. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν θα σχολιάσω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μπόνη γιατί συμμερίζομαι τα περισσότερα από αυτά που είπε. Θέλω να συγχαρώ πάντως τον ομιλητή για την παρουσίαση την οποία έκανε για τη δουλειά την οποία έχει ολοκληρώσει και για τον τρόπο με τον οποίο παρουσίασε την έκθεσή του. Το έκανε με συνθετικό τρόπο, εξέφρασε τις πέντε βασικές ανησυχίες και αναφέρθηκε και στις αναχώρα εκθέσεις, οι οποίες ολοκληρώθηκαν για πρώτη χρονιά περιγράφησαν με πάρα πολύ σωστό τρόπο και περιλαμβάνουν πάρα πολλές χρήσιμες κυρίως πληροφορίες και ε, εγώ βλέπω και την αντίστοιχη για τη χώρα μου. Όπως έλεγε ο συνάδελφος Μπόνι, έχουμε να κάνουμε με κάποιες τάσεις τις οποίες μας παρουσίασε ο Διευθυντής της Εξωτερικής Υπηρεσίας είναι μερικές φορές τα στοιχεία αυτά θα έλεγα σοκαριστικά ε, για, ιδιαίτερα για την χρήση των ναρκωτικών στα σοφρονιστικά ιδρύματα. Πώς σε ένα κλειστό ίδρυμα μπορεί να κυκλοφορούν τέτοιου είδους ουσίες. Το θέμα βέβαια εδώ είναι περισσότερο εθνικό παρά ευρωπαϊκό η Επιτροπή μας στα πλαίσια της αξιολόγησης του σοφρονιστικού συστήματος θα πρέπει να προσπαθήσει να δει σε τι οφείλεται η κατάσταση αυτή. Καταρχάς, τίθεται το θέμα των, της αύξησης των θανάτων από υπερβολική δόση. Ε, το παρατηρητήριο πώς αντιδρά και πώς εξηγεί αυτή την κατάσταση υπήρξε μια αύξηση της κατανάλωσης των πιο επικίνδυνων ουσιών, ε, παρεσθητικών σαν παραδείγμα. Υπήρξε μια αποτυχία θα έλεγα των μέτρων αντιπαράθεσης ε, με το λαθρεμπόριο ή υπήρξε μια μεγάλη αύξηση της κατανάλωσης. Πώς εξηγεί λοιπόν το παρατηρητήριο την αύξηση των θανάτων από υπερβολική δόση. Μια άλλη ερώτηση που δεν έχει άμεση σχέση με την έκθεση αυτή, αλλά είναι μια ερώτηση που νομίζω παρουσιάζει ενδιαφέρον. Ο Επίτροπος Αβραμόπουλος αναφέρθηκε στην τεράστια οικονομική αξία την οποία εκπροσωπεί το λαθρεμπόριο των ναρκωτικών. Είναι τρομακτικό το ύψος και ίσως και αυτό αποτελεί και το βασικό κίνητρο. Το εύκολο κέρδος λοιπόν είναι αυτό το οποίο ε, θα έλεγα ενισχύει την ε, δραστηριότητα αυτή την παράνομη και στη συνέχεια την αύξηση ε, των εξαρτημένων από τις ουσίες αυτές. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι καλές πρακτικές σε διάφορες χώρες που μπορεί να υιοθετηθούν στο σύνολο της Ένωσης για να αντιστρέψουμε λίγο την τάση. Ο κύριος Χωστέλε, ευχαριστώ πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μπεν και τον κύριο Κοέλιο για τις ερωτήσεις θα σας ε, απαντήσω προσπαθώντας να μην σας κάνω μια δεύτερη παρουσίαση. Αν θέλετε επιπλέον στοιχεία, ξέρετε που μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Το πρώτο που είχα να πω για το σχόλιο, για την ε, κοκαίνη και την αυξή της ευθεσιμότητας. Καταρχάς, σας είπα ότι έχουμε μία ομάδα διαφορετικών δικτών που φαίνεται ότι καταδεικνύει ότι υπάρχει πιο πολύ κοκαίνη στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν έχουμε ακόμα οποιαδήποτε ένδειξη για αύξηση των ε, πελατών, των καταναλωτών. Γι' αυτό σας είπα ότι παρακολουθούμε την κατάσταση προσεκτικά. Τώρα, σε σχέση με αυτό και μιλήσατε για την ε, αστυνομία, τα σώματα επιβολής του νόμου, τη Γεροπόλ. Καταρχάς υπάρχει στην συνεργασία η Γεροπόλ ήταν και η πρώτη υπηρεσία που, την οποία επίσημα επισκέφθηκα από την ανάληψη των καθηκόντων μου. Προετοιμάζουμε μια ενημέρωση του Μνημονίου Συνεργασίας και μαζί με τη γεροπόλα συνεργαστήκαμε και πριν από τρεις εβδομάδες η γεροπόλα παρουσίασε τη 8 την έκθεση για την αξιολόγηση των απειλών και του κινδύνου. Υπάρχει στι 8 στην έκθεση αυτή ένα ιδιαίτερο τμήμα το οποίο είναι αφιερωμένο στα ναρκωτικά και έχουμε και την έκθεση για την ιστορική ε, αγορά. Και αυτό από κοινού με την καταρτίστηκε και από τις πληροφορίες που λάβαμε και που παρουσιάστηκαν στο ΚΟΖΗ στο Συμβούλιο, τις πληροφορίε που έχω εγώ στην διάθεσή μου, είπα περιπτώσει, ενημερωθήκαμε ότι θα υπάρχει μία και όχι δύο προτεραιότητες πλέον για τα ναρκωτικά, αλλά θα περιλαμβάνει όλα τα ναρκωτικά αυτή τη φορά. Όλες τις ουσίες. Για να εξασφαλίσουμε ότι όταν τα κρατημέλη ακολουθήσουν την ε, σύσταση αυτή, όλα τα ναρκωτικά θα βρίσκονται στον ίδιο βαθμό προτεραιότητας, γιατί όλα περιλαμβάνονται από την προτεραιότητα αυτή. Αυτό το, ήταν το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο τώρα για τις νέες ψυχοτρόπες ουσίες. Νομίζω ότι μία από τις βελτιώσεις της νέας νομοθεσίας όταν το καλό εφαρμοστούν είναι ότι θα περιορίσουν και το χρόνο εφαρμογής ε, των μέτρων από πλευρά των κρατών μελών όταν αυτά αποφασιστούν από 12 σε 6 μήνες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα υπάρξει η απόφαση να υπάρξει έλεγχος. Ε. Θα μειωθεί σημαντικά ο χρόνος από την ε, απόφαση μέχρι την υλοποίηση της απόφασης και κάτι άλλο που ήδη προβλεπόταν από την κοινή δράση των 97 ήδη. Μας είπατε τι, σημα... τι χρειάζεται το ESDD για να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Η απάντηση είναι αρκετά απλή βραχυπρόθεσμα. Εμείς και οι εταίροι μας εργαζόμαστε από αυτού για τον προπολογισμό για το 2017. Υπήρξε και μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπάρξει επιπλέον προϋπολογισμός για την βάση δεδομένων του EDFT που αποτελεί το βασικό εργαλείο μας. Θα χρειαστεί λοιπόν αυτό για δύο-τρία χρόνια για να βελτιώσουμε το εργαλείο αυτό. για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην αύξηση των παραχόμενων ναρκωτικών. Θα υπάρξει λοιπόν αυτή η αύξηση. Έχουμε λοιπόν τους πόρους που χρειάζονται βράχη πρόθεσμα, μα μέσω πρόθεσμα θα ήμουν πιο προβληματισμένος, όχι απαραίτητα Ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν θα είμαστε ασφαλώς η μοναδική υπηρεσία που το λέει αυτό, αλλά χρειαζόμαστε ένα όραμα για να δούμε ποια θα είναι η πραγματικότητα και ποιος θα είναι ο ρόλος μας στην Ευρώπη μετά το Brexit. Γιατί το Brexit σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που θα έχει στη χρηματοδότηση και στον προπολογισμό ενδεχομένω και κατά πάσα πιθανότητα θα έχει τεράστιο αντίκτυπο για όλες τις υπηρεσίες, όλες τις εξωτερικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα αυτές του κλάδου μας. Η τελευταία σας ερώτηση έχει να κάνει με την στρατηγική της ε, EMCDDA. Με χαρά να σας δώσω, Πρόεδρε, το φλάδι αυτό. Είμαστε στα μέσα της υλοποίησης για το φετινό έτος και θα πρέπει να γίνει κάποια, να ολοκληρωθεί ένα διοργάνωση η οποία ξεκίνησε. Να περάσω στον κύριο Κοέλιο να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη θετικά σας σχόλια και για τη συνεχιζόμενη υποστηρίξή σας. Χαίρομαι ιδιαίτερως που σας αρέσει αυτή η έκθεση αναχώρα, ιδιαίτερα γιατί πρόκειται για ένα παράδειγμα διαφορετική συνεργασία και διαφορετική εργασία στο πλαίσιο αυτό. Έχουμε 6-7 συναδέλφου από διαφορετικέ υπηρεσίε που ήταν πάρα πολύ παραγωγικοί και επικοδομητικοί και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτού. Σκοπό είναι να επικεντρωθούμε πιο πολύ στου πελάτε μα και εσεί είστε ένα από του βασικού μα πελάτε. Χαίρομαι λοιπόν που βρίσκεται τι πληροφορίες αυτές εμ, οι πληροφορίε για τι φυλακέ συμφωνώ ότι προκαλούν σοκ ομολογουμένω και καταλαβαίνω φυσικά την είναι πιο πολύ αρμοδιότητα των κρατών μελών, δεν λέω, και όχι τόσο πολύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να σα πω ότι πρόκειται για ένα γενικό ζήτημα. Και γι' αυτό τα θέματα που από τον των ναρκωτικών, τη ριζοσπαστικοποίηση στι φυλακέ. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι οριζόντια, εγκάρσια και όλα σημαίνουν ότι θα πρέπει να επενδύσουμε κόπο και πόρους στις φυλακές. Προφανώς δεν υπάρχουν σαφείς ε, λύσεις. Θα πρέπει να αφιερωθεί πιο πολύ χρόνος, πιο πολύ πόροι από πλευράς EMCDDA. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή των προγραμμάτων και τις πρωτοβουλίες σε ό,τι αφορά το EMPS τώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να το αναφέρουμε το γεγονός ότι αυτή η νέα συμφετική κάναβης είναι τόσο συμπυκνωμένη και κατά συνέπεια μικρότερη σε όγκο, δυσκολεύει την, ε, τον έλεγχο στα σαφρονιστικά ευρέματα. Τελευταίο ερώτημα, τελευταία παρατηρήση που κάνετε για τις ε, υπερβολικές δόσεις. Για τις υπερβολικές ε, δόσεις, τα περιστατικά αυτά υπερβολικές δόσεις, ξέρουμε ότι κάποιες από τις αλλαγές έχουν να κάνουν και ε, με αλλαγή των στοιχείων και βελτίωση της καταμέτρησης και των στοιχείων καταμέτρησης. Μιλάμε για νέα συνθετικά ήδη. Αλλά δεν καταχωρίζονται όλα από κάθε εργαστήριο με τον ίδιο τρόπο. Άρα όλο αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το παρακολουθούμε. Ύστερα, το γεγονός ότι υπάρχουν ε, αναμίξεις, μείγματα και ότι ο κόσμος ε, τα χρησιμοποιεί παίζει και αυτό σημαντικό ρόλο. Και ύστερα το γεγονό ότι έχουμε πιο πολλέ. ότι υπάρχουν πιο πολλές φεντανίλες και αυτό φυσικά επηρεάζει τα στοιχεία. Τώρα, για αυτούς που χάνουν τη ζωή τους λόγω προβολικής δόση, ε, ενώ χρησιμοποιούν μεθαδόν, για παράδειγμα, ιατρικές ε, ουσίες, ε, στις πιο πολλές περιπτώσεις, αν όχι σε όλες, δεν βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Καταρχάς, λοιπόν, θα πρέπει να βελτιώσουμε την παρακολούθηση, αλλά ένας παράγοντας είναι και αυτός, ότι δεν είμαστε ακόμα απόλυτα καλυμμένοι μόνο 15%. 50% ε, συγγνώμη. Κάποιες χώρες ήταν στο 20%. Υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά δεν, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Μιλάμε για 24 δισεκατομμύρια από 25 έως 31 εκατομμύρια. Τώρα, πέρσι, και το ανέφερε και ο Επίτροπος Αβραμόπουλος, είναι σημαντικό το στοιχείο αυτό. Ακόμα και αν δεν βλέπουμε τον κόσμο να χάνει τη ζωή του στους δρόμους ε, λόγω χρήσης ναρκωτικών, εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό τμήμα της αγοράς ε. και λόγω του οργανωμένου εγκλήματος. Προσπαθούμε λοιπόν να αναδιοργανώσουμε τα στοιχεία και τα επόμενα χρόνια θα υποβάλουμε πιο ακριβή αριθμητικά στοιχεία. Για τη νέα λοιπόν έκδοση της αξιολόγησης το 2019 αναμένεται ότι θα έχουμε καινούργια στοιχεία στη διάθεσή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση και για την έκθεση και για τη στρατηγική αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον κύριο Κοέλιο και τον κύριο Μπόνη. Και συνάδελφοι, να περάσουμε στο σημείο 16. Είναι εδώ και οι προσκεκλημένοι μας. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ που έχετε καταφτάσει στην ώρα σας. Μία παρουσίαση από τον κύριο Ναβαρέτε από την Europol. the colleagues, Europol has been producing the annual EU Terrorism Situation and Trend Report, TSAT, since 2007. Η έκθεση αυτή λοιπόν μας παρουσιάζει συνολικά μια περιγραφή του τρομοκρατικού φαινομένου κύριος Μανουέλ Ναβαρέτε από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, του, από το κέντρο το Ευρωπαϊκό για την Καταπολέμηση της Τρομοκρατίας και την Ευρωπόλ. Ήταν μια μεγάλη εβδομάδα, είναι πέμπτη απόγευμα. θα μου ζητήσετε να διακόψουμε για πέντε λεπτά, γιατί ίσως να υπάρχει μια σύγχυση με το timing, με το χρόνο. Αν δεν σας πειράζει να περιμένετε λοιπόν λίγο. Πέντε λεπτά διακοπή.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 I'd like to welcome the EPP coordinator to her seat. Um, with all respect, now that I'm on the microphone, thank you, Roberta, for your presence. Ευχαριστώ, Ρομπέρτα, για την παρουσία σου εδώ. Libe is meeting almost every week, unlike... Εμείς συναντώμεθα κάθε εβδομάδα, όχι σαν άλλες επιτροπές που το κάνουν μια φορά το μήνα σχεδόν και γι' αυτό υπάρχουν πολλές απουσίες. Αλλά πάντως αναμεταδίδεται δικτυακά η συνεδρίαση. Βλέπω εδώ και την συντονίστρια και ε, πραγματικά μίζω μέλος της Επιτροπής μας ε, που ήρθε. Την ποιότητα την έχουμε, ποσότητα δεν έχουμε. Μη με κοροϊδεύετε, ε, πιέζομαι κι εγώ. Η αλήθεια είναι ότι όταν ο κόσμος αρχίζει και γελάει μαζί σου, είναι η στιγμή μάλλον που πρέπει να φύγει κανείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έτσι κι αλλιώ έχουμε χρόνο, κανονικά τώρα θα αρχίζαμε την συγκεκριμένη συζήτηση. Um, welcome again Mr. Um, head of the European at Europol. Λοιπόν, είναι ο υπεύθυνο για τα θέματα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Ευρωπόλ. Έχουμε επαφές με την Ευρωπόλ πρόσφατα. Επαφές είναι τακτικές, έχουν οριμάσει σε σχέση με το τι ίσχυε πριν μερικά χρόνια. Ε, ευχαριστώ και τους παρόντες, τις παρούσες μάλλον συναδέλφους. Ξέρω ότι ε, μια, υπήρξε μια πάρα πολύ εντατική εβδομάδα, απαιτητική εβδομάδα και σας ευχαριστώ που είστε παρούσες εδώ. Λοιπόν, ο κύριος Ναβαρέτ θα είναι σύντομος, θα μας μεταφέρει όμως τα βασικά σημεία. Δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση ήδη από το, για το και παρουσιάζει γενικά την κατάσταση του φαινομένου της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριος Ναβαρέτ, σας καλωσορίζω. Είναι υπεύθυνο για τα θέματα λοιπόν καταπολέμησης της τρομοκρατίας στην Οροπόλ. Καλώς ήρθατε και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας καλησπερίζω όλους και όσους μας παρακολουθούν διαδικτυακά. Είμαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω την έκθεση του 17 που αναφέρεται στα στοιχεία και στα δεδομένα από το 16 βέβαια. Η έκθεση το TISAT λοιπόν 17 είναι δύο χρόνια που λειτουργεί το TISAT και μαζί με τα διάφορα μέλη αξιολογούμε τα δεδομένα, αξιολογούμε τους αριθμούς που έχουμε και τα καταθέτουμε συγκεντρωτικά. Θα περιμένατε από πλευράς μας περισσότερα, κάτι περισσότερο από ορισμένα στοιχεία αριθμητικά και ποσοτικά. Και γι' αυτό μπορώ να σας παρουσιάσω λίγο μια αξιολόγηση του πώς πάει η κατάσταση σήμερα, το πώς επηρεάζει την καθημερινότητα των πολιτών μας, πώς προχωρούμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, πώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Europol και κυρίως τα κράτη-μέλη αντιμετώπισαν το θέμα αυτό το 2016 και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία που ήδη έχουμε μέχρι τώρα ζητήθηκε από την υπηρεσία μας, από την Προεδρία, να προετοιμάζει μια εξαμηνία έκθεση για τις εξελίξεις στην τρομοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας παρουσιάσουμε κάποια από τα ευρήματα της έκθεσης αυτής, την οποία εμείς ε, ε, προετοιμάζουμε και για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Βλέπετε ότι το 2016 ένα σύνολο 142 αποτυχημένων και ε, υπήρξαν βάση περιπτώσει απόπειρες οι οποίες ε, δεν ολοκληρώθηκαν, όμως 142 θύματα πέθαναν στις ε, επιθέσεις αυτές και τραυματίστηκαν 379 άτομα. Οι αριθμοί είναι λίγο καλύτεροι από το 2015. Υπάρχει μείωση των θυμάτων Υπάρχει ε, μείωση των επιθέσεων για λόγους που θα σας εξηγήσω σύντομα. Αλλά παρότι έχει υπάρξει βελτίωση σχετικά με τον προηγούμενο χρόνο, η εικόνα είναι ότι η απειλή παραμένει ιδιαίτερα υψηλή και δεν ήταν καθόλου καλή χρονιά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις. Η επιλογή των στόχων γίνεται με διαφορετικό τρόπο συγκεντρώνουν την προσοχή του τώρα σε μεγάλες συγκεντρώσεις πολιτών. Χρησιμοποιούν ε, διάφορες μορφές παγίδευσης με εκρηκτικά και ε, αυτοί οι οποίοι διαπράττουν την απόπειρα δεν είναι και τόσο οργανωσμένοι, εμπνέονται από ε, άλλες τρομοκρατικές ενέργειες. national venue or close Κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό λειτουργεί πολλαπλασιαστικά ε, και προκαλεί την προσοχή των μέσων ενημέρωσης. Το 2015 όμως είδαμε ότι είχαμε πολύ περισσότερα θύματα από ότι το 2016 αλλά όπως είπα η αντίληψη της απειλής είναι υψηλότατη. Η μείωση οφείλεται στο ότι οι επιθέσεις εξτρεμιστικών ακραίων εθνικιστικών ή υπερεθνικιστικών ομάδων μειώθηκαν. 374 θύματα από τα 379 οφείλεται λοιπόν σε τέτοιου είδους επιθέσεις και όλοι, όλα τα θύματα που έχασαν τη ζωή τους οφείλονται στις επιθέσεις αυτές. Οι, οι επιθέσεις των ζιχαντιστών αυξήθηκαν το 2016 Γίνονται προσπάθειες ε, που ενισχύονται και από την ε, ε, Europol. Οι περισσότερες από τις απόπειρες αυτές έγιναν στην Γαλλία, μετά στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Αυστρία και την Ιταλία. Υπήρξαν λοιπόν δράσεις ε, εις βάρος των τρομοκρατικών ομάδων σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν 13 ε, επιθέσεις που οφείλονται στις λεγόμενες θρησκευτικού τύπου ένοπλες ομάδες. Η πιο πρόσφατη ήταν στις 22 Μαρτίου στις Βρυξέλλες, ε, χάθηκαν 30 πολίτες στις 4 Ιουλίου στη Νίκαια, όπου σκοτώθηκαν 85 πολίτες και στις 19 Βερολίνου στο Βερολίνο με 16 θύματα τουρίστες και ε, Γερμανούς πολίτες. Έγιναν όμως επιθέσεις και στην Τουρκία και στην Αίγυπτο, στο Μαλί, την Αλγερία, τον Ήγυρα, το Αφγανιστάν, τον Μπαγκλαντές και την Ινδονησία και υπήρξαν και εκεί θύματα Ευρωπαίοι, είτε έχασαν τη ζωή τους είτε τραυματίστηκαν. Υπήρξαν επίσης και απαγωγές πολιτών της Ένωσης εκτός Ευρώπης. Οι τρομοκράτες θεωρούν ότι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των δυτικών χωρών είναι υψηλής ποιότητας στόχος, έτσι ώστε να εισπράξουν τα λίτρα. Το 2016 το ποσοστό των απαχθέντων ήταν ιδιαίτερα υψηλό, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος. Λιβύη, Μαλή και Φιλιππίνες. Θεωρούμε ότι οι ένοπλες τρομοκρατικές ομάδες δεν επιλέγουν πολίτες μιας συγκεκριμένης εθνικότητας, αλλά με οπορτουνιστικό τρόπο αναζητούν τα θύματα τους. Τώρα, πώς έχει η κατάσταση της τρομοκρατίας σήμερα. Η κατάσταση δυστυχώς είναι ρευστή, πιο ρευστή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει σωστά προγραμματισμένες επιθέσεις από δίκτυα τρομοκρατικών ομάδων με μαχητές οι οποίοι προέρχονται είτε εκτός Ευρώπης αλλά και θόρμητες επιθέσεις που γίνονται από μεμονωμένους δράστες ε, και πολλές φορές προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν την υπηκότητα ή άδεια παραμονής εδώ και πολλά χρόνια στην Ένωση. Νίκαια, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκόλμη. Ε, οι ξένοι μαχητές στις περισσότερες περιπτώσεις παραμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν παραμείνει στην Ένωση για αρκετά χρόνια. Οι δράστες μπορεί να ελέγχονται άμεσα από το Ισλαμικό κράτος ή μπορεί να εμπνέονται από τη ρητορική και την ιδεολογία. Δεν είναι προφανής η σχέση τους με το Ισλαμικό κράτος, φαίνεται όμως ότι εμπνέονται όπως είπα και από τον τρόπο λειτουργίας επηρεάζονται από την προπαγάνδα του ISIS έτσι ώστε οι δράστες να εμφανίζονται σαν στρατιώτες του Χαλιφάτου, ακόμα και αν δεν έχουν σχέσεις μαζί του. Πολλοί δράστες ήταν γνωστοί στην αστυνομία και είναι πολύ δύσκολο να γνωρίζει κανείς το επίπεδο κινδύνου που αντιπροσωπεύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ε, δεν είχαν θεωρηθεί άμεσος κίνδυνος, πάντως πολλοί από αυτούς είχαν και ποινικά προηγούμενα, μητρώα, αλλά δεν είχαν σχέση με την τρομοκρατία. Εδώ βλέπουμε τους ε, αριθμούς, δεν βλέπουμε δηλαδή. Υπήρξε μείωση ε, μαχητών, του αριθμού των μαχητών που πηγαίνουν στη Λιβύη και κυρίως στη Συρία για να πολεμήσουν ε, κανονικά ο αριθμός έπρεπε να αυξηθεί, αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες βλέπουν ότι ε, δεν έχουν υπάρξει και επιστροφές ιδιαίτερα υψηλές από τις χώρες αυτές και αυτοί που επιστρέφουν είναι συνήθως ανήλικοι και γυναίκες. Τώρα ποιοι είναι οι τρομοκράτες. Έχουμε διαφορετικά προφίλ. Κάποιοι επιστρέφουν από την περιοχή, από τις εμπόλεμες περιοχές, κάποιοι δεν έχουν φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κάποιοι ε, λειτουργούν ε, υπηρετώντα ε, τον ISIS. Βλέπουμε αύξηση του αριθμού γυναικών οι οποίες ενθαρρύνουν την διάπραξη των τρομοκρατικών ενεργειών. Οι ξένοι μαχητές σήμερα ριζοσπαστικοποιούνται πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι ξένοι μαχητές κινητοποιούνται όχι μόνο για θρησκευτικούς λόγους, Πολλές φορές υπάρχουν διαφορετικά στοιχεία, οικογενειακή πίεση, το λεγόμενο peer pressure, δηλαδή εξωθούνται από τους ομοίους τους να προβούν σε τέτοιου είδους πράξεις. Τι όπλα χρησιμοποιούν. Χρησιμοποιούν αρκετά προχωρημένα όπλα, όπως είδαμε στο Παρίσι και στις Βρυξέλλες, και κάποια τυχαία όπλα, μερικές φορές, όπως ε, μαχαίρια και οχήματα με τα οποία χτυπούν τους ε, αθώους ε, πολίτες. Εδώ φαίνεται ο ρόλος της προπαγάνδας τον οποίο, την οποία χρησιμοποιεί η Αλκάιντα. Είναι βασικό κομμάτι της στρατηγικής των τρομοκρατών προωθούν την επικοινωνία, τη βία, ε, όπως επίσης και συλλέγουν έσοδα. Στόχος της προπαγάνδας το 15 και μετά το 2015 έχει αυξηθεί. Υπάρχει θα έλεγα αυξημένη ε, προπαγανδιστική δραστηριότητα. ανακυκλώνουν την προπαγάνδα, την παλαιά, διότι δεν παράγονται εύκολα νέα, φιλμ και βίντεο ο αριθμός των νέων βίντεο που παράγεται από το Ισλαμικό κράτος μειούται. Τα μηνύματα έχουν περάσει από τα συνθήματα για τον νικηφόρο Ισλάμ σε εκκλήσεις για επιθέσεις εκδίκησης και αντεκδίκησης. Στην ουσία έχουν περάσει από την επιτυχία στην αποτυχία. Also, Al-Qaeda is using Παρ' όλα αυτά λοιπόν, αν συγκρίνουμε το τι γινόταν πριν μερικά χρόνια, βρίσκονται σε χαμηλό επίπεδο. Εμείς προσπαθήσαμε στο εσωτερικό της υπηρεσίας μας να δημιουργήσουμε νέες μονάδες συλλογής περιεχομένου παρεμβαίνουμε στο διαδίκτυο ζητώντας από αυτούς οι οποίοι παρέχουν φιλοξενία σε τέτοιο είδους ε, υλικό να το αποσύρουν. Συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη και επίσης κάνουμε προσπάθειες ε, ε, για να απομακρύνουμε και να μετριάσουμε την διάδοση των προπαγανδιστικών δραστηριοτήτων στο διαδίκτυο. Έχουμε δημιουργήσει και ένα εσωτερικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση φόρουμ για αυτό το λόγο. Το τι θα γίνει στο μέλλον είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαντέψει κανείς. Είναι όμως σαφές ότι η κατάσταση την οποία έχουμε, έχουμε μπροστά μας γίνεται ασταθέστερη και ως εκ τούτου μη προβλέψιμη. Περιμένουμε από τους τρομοκράτες να συγκεντρωθούν σε συγκεκριμένους στόχους, αλλά επίσης και αδιάκριτα να προβαίνουν σε δολοφονίες. Το είδαμε αυτό στις αρχές του 2017. Τα τελευταία χρόνια είδαμε τρεις τύπους στόχων. Καταρχάς, ο ένας στόχος είναι αδιάκριτες επιθέσεις, Δεύτερον, συμβολικά για τον τρόπο ζωής της Δύσης σημεία. Και τρίτον, εκπρόσωποι αρχών και κυρίως αστυνομία. Πώς τώρα η κατάσταση στο Ιράκ και στη Συρία θα επηρεάσει την κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος. νομίζουμε ότι όταν ιτηθεί το Ισλαμικό κράτος από τις δυνάμεις του συνασπισμού στη Συρία, τότε οι μαχητές θα προσπαθήσουν να δράσουν με διαφορετικό τρόπο. Πρώτον θα συνεχίσουν να κάνουν αντάρτικο πια στην περιοχή έως ότου εξοντωθούν από τους εχθρούς τους. Δεύτερον θα παραμείνουν δραστήριοι στη Συρία και στο Ιράκ αλλά σε ε, παράνομες μορφές δράσης. Και τρίτον, ίσως να παραμείνουν σε ορισμένους θυλάκους τους οποίους ίσως να μπορέσουν να κρατήσουν μετά την ήττα τους. Κάποιοι επίσης θα καταφύγουν και σε γειτονικές χώρες και κάποιοι θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα οι ξένοι μαχητές. Τώρα, ανεξάρτητα της επιλογής που θα κάνουν, θα παραμείνουν απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οργάνωση παραμένει, ε, θα έλεγα, επικίνδυνη, το, η Αλκάιδα και το Χαλιφάτο έδειξαν από το 2015 και μετά ότι είναι ικανές να, να επιτεθούν σε πάρα πολλά σημεία της Ένωσης. Η εικόνα την οποία έχουμε λοιπόν για το 2017 είναι παρόμοια με του 16. Οκτώ επιθέσεις τους πρώτους... Ε, Θα ήθελα με την ευκαιρία των παρατηρήσεων μου να αποτίσω φόρο τιμή στην εργασία που έχουν κάνει ε, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πολυμερής ε, συνεργασία έχει σώσει πολλές ζωές. Και το ξαναλέω και το τονίζω, έχει σώσει πολλές ζωές. Ο ρόλος ε, της ε, Ευρωπόλ είναι να υπηρετήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο ε, την Ευρώπη. Έχουμε δευτερογενείς ομάδες, έχουμε ικανότητες ανάλυσης. Οι γνώσεις μας, οι εμπειρίες μας είναι ακριβώς στην υπηρεσία της Ευρώπης οι 28 χώρες μέλη και οι 11 επιπλέον χώρες συμμετέχουν στο σύστημα της ε, Europol και μέχρι το Μάιο του 2017 ε, είχαμε 7.250 ε, πράξεις. Έχουμε περίπου 8.500 ε, ε, ε, ξένους μαχητές ταυτοποιημένους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά στοιχεία που αφορούν μονάχα 12 μήνες. Επιπροσθέτως, τα κράτη-μέλη τώρα χρησιμοποιούν εντατικότερα το σύστημα πληροφοριών της Europol. Μέχρι τις 11 Μαΐου του 2017 τα κράτη-μέλη είχαν κάνει παραπάνω από 600.000 έρευνες ε, στο σύστημα της ε, Ευρωπόλ. Δηλαδή χρησιμοποιείται καθαρά το σύστημα αυτό όσον αφορά τις, ε, τις επιχειρήσεις τρίτων μερών και αυτές βοηθούν πάρα πολύ έτσι ώστε να εξουδετερώνονται οι τρομοκράτες πριν προλάβουν να κάνουν κακό εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και συνεργαζόμαστε με το FBI και παίρνουμε πληροφορίες ε, δηλαδή ε, από το FBI των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες από διάφορες πηγές, κυρίως για τους ξένους μαχητές, έτσι ώστε να κάνουμε καλύτερα την ερευνητική δουλειά. Europol supported, I have my figures here, Κάπου είχα τα, τα στοιχεία μου, αλλά που τα βάλα, λέει ο μιλητής, δεν ξέρω. Here we are. 137 έρευνες ε, έγιναν το 2016, περίπου 50% αύξηση σε σχέση με το 2015. Έχουμε τώρα από 30 ε, χώρες ε, και ε, ε, συμβαλόμενα μέρη, εκπροσώπου CT, η Internal Referral Unit έχει στείλει περίπου 30.000 ε, υπηρεσίες πληροφορίας και σε 84% των περιπτώσεων έχουμε Έχουμε ανταποκριθεί στο αίτημα ε, το, το οποίο μας έχει ε, γίνει. Σε συνεργασία με την Κομισιόν έχουμε ξεκινήσει το Internet Forum, αυτήν την ε, ε, πρωτοβουλία έτσι ώστε να μειώσουμε την προσβασιμότητα των τρομοκρατών σε περιεχόμενο ε, και επίσης ε, για να δημιουργήσουμε αναλυτικές δυνατότητες στην επιγραμμική πληροφόρηση. Επίσης, εδώ και ένα χρόνο περίπου έχουμε και μια ομάδα η οποία παρακολουθεί επιγραμμικά όλες τις προπαγανδιστικές προσπάθειες συνεργαζόμαστε με εμπειρογνώμονες της τρομοκρατίας ε, για περιπτώσεις ε, κατά χρηστικής ε, εκμετάλλευσης παιδιών και προπαγάνδας online. Βεβαίως τώρα επικεντρωνόμαστε και στις χώρες των Δυτικών ε, Βαλκανίων και κυρίως θέλουμε να διατηρήσουμε το υψηλό επίπεδο συνεργασίας ε, που ξεκινήσαμε τους τελευταίους μήνες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τις αρχικές μου παρατηρήσεις ε, θα ήθελα να τις ολοκληρώσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα μέλη του. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίες και κύριοι βουλευτές για την αποφασιστικότητα με την οποία αντιμετωπίζετε τα θέματα αυτά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε όσο καλύτερα γίνεται τη δουλειά μας εμείς οι εκπρόσωποι των αρχών επιβολής ε, του νόμου και της, ε, ε, των υπηρεσιών πληροφοριών αλλά και εσείς πρέπει να κάνετε την δουλειά σας και την κάνετε είδαμε ότι το 2016 είχαμε αύξηση των, ε, μείωση συγγνώμη, των θυμάτων, αλλά αυτό δεν αρκεί. Και ένα να είναι το θύμα είναι ένα παραπάνω από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεσμεύομαι και δεσμεύομαι και το της ε, Europol ε, να υπερπροσπαθήσουμε έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις προκλήσεις. Είναι δύσκολο αυτή την ώρα να δει κανείς το φως στην άκρη του τούνελ, γιατί τώρα είμαστε στο, στην ε, ε, μέση του τούνελ. Εγώ ξέρω τι σημαίνει τρομοκρατία. Εγώ για πάρα πολλά χρόνια ε, πολέμησα την οργάνωση ΕΤΑ και ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει. Και ξέρω όμως ότι υπάρχει δρόμος για να βγούμε από το τούνελ και υπάρχει και ζωή μετά το τούνελ και αυτή η ζωή έχει ένα όνομα, λέγεται δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω για όποιες ερωτήσεις έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ναβαρέτη και είδατε ότι όσο μιλούσατε ήρθαν και άλλα μέλη στην αίθουσα και βεβαίως συμφωνούμε με τα όσα μας είπατε. Και εμείς συζητούμε πώς ε, μπορούν να ενδυναμωθούν ε, και μάλιστα με έντονο τρόπο οι σχέσεις ανάμεσα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και την Europol. Συμφωνούμε λοιπόν μαζί σας ε, ε, ότι είναι σημαντικές οι επιχειρήσεις, ε, είναι γεγονός ότι δεν μπορούν να δημοσιοποιούνται όλες οι επιχειρήσεις, αλλά υπάρχουν. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Δύο δικές μου ερωτήσεις. Η έκθεση Τσέν. Υπάρχουν καλοί ε, δημοσιογράφοι οι οποίοι μας ε, δίνουν και πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις, σχετικά με το τι σημαίνει με την, συμβαίνει με την οργάνωση Ισλαμικό κράτος, σχετικά με τις ομότητες οι οποίες ε, λαμβάνουν χώρα, αποκεφαλισμοί, χρήση μαχαιριών κτλ. Παγιδευμένα αυτοκίνητα. Το ζήτημα είναι και φαντάζομαι ότι και το γνωρίζουν και οι αναλυτές της Europol. Ποια είναι η ε, προστιθέμενη πληροφορία που δεν γνωρίζουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι αναλυτές πληροφοριών λένε ότι ίσως υπήρξε αύξηση λόγω του Ραμαζανιού, αύξηση των επιθέσεων, λόγω του, των του Ραμαζανιού ή απλώς ε, γιατί υπήρχαν, ε, ε, κάνανε άνθρωποι ψυχοτικά επεισόδια, δεν ξέρουμε ακόμα. Πρέπει να γίνει μια ανάλυση. Και το λέω αυτό γιατί εδώ δεν μιλάμε μονάχα για τις απώλειες των συγκεκριμένων ανθρώπινων ζώων. Μιλάμε για τη γενικότερη σκιά της τρομοκρατίας στην δημοκρατία, στην ζωή μας κλπ. Επομένως θα πρέπει να γίνει κάποια ανάλυση ε, ε, ε, ε του τρόπου πληροφόρησης, του τρόπου με τον οποίο θα πρέπει να χειρίζονται την πληροφορία ή τα μέσα ενημέρωσης. Πού βρίσκεται η αλήθεια πίσω από όλα αυτά. Το δεύτερο ζήτημα είναι το θέμα του ίντερνετ, του διαδικτύου. Χρειαζόμαστε και το facebook, χρειαζόμαστε και γιατί βρίσκουμε υλικό εκεί. Ποιε είναι οι τελευταίες εξελίξεις και οι απόψεις σχετικά με αυτά τα δίκτυα και το ίντερνετ. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχει έξαρση στη διάρκεια των εκλογικών, προεκλογικών ε, διαδικασιών. Ε, λοιπόν, θα ξεκινήσουμε πρώτα με την Ανταλή Βίσπακ. <laughs> Ε. Σας κάνω εντύπωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να ευχαριστήσω και για την παρουσίαση αυτή, η οποία ήταν πραγματικά πολύ συνοπτική, παρά το γεγονό ότι δεν καταφέραμε να διαβάσουμε το έγγραφο πριν από την παρουσίαση. Δυστυχώ δεν δημοσιεύτηκε εξ αρχή, αλλά σε κάθε περίπτωση εξετάζεται την ετήσια έκθεση, η οποία μα επιτρέπει να δούμε και το μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρά το γεγονός ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις έχουν την τάση να πολλαπλασιάζονται. Θεωρούμε ότι η έκθεση αυτή αποτελεί μια πολύ σημαντική βάση για μας που καλούμαστε συχνά να νομοθετήσουμε για το θέμα αυτό, το οποίο προφανώ επηρεάζει τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Αναλύσεις, αξιολογήσεις ε, των απειλών, του τρόπου λειτουργία, όπως ε, αναφέρατε σε διάφορες περιστάσεις, ε, τη φύση των τρομοκρατικών επιθέσεων. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά δεδομένα σε ό,τι αφορά τη δουλειά που έχουμε να κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην ε, παρουσίαση μιλήσατε για διάφορους ε, τύπους, προφίλ ε, τρομοκρατών που εμπλέκονται σε τρομοκρατικές δράσεις. Υπάρχουν ανάλυσεις, πληροφορίες τις οποίες θα μπορούσατε να δημοσιεύσετε και θα μας επέτρεπαν ενδεχομένω να βελτιώσουμε το σκέλος της πρόληψης, πρόληψης της ε, ταυτοποίησης των ε, ενδεχομένων τρομοκρατών. Είπατε ότι η κατάσταση προφανώς ε, προκαλεί έντονα συναισθήματα, αλλά πώς μπορούμε να εντοπίσουμε κάποια προφίλ. Εγώ είμαι Γαλλίδα και προχθές το άτομο το οποίο έδρασε στην Τροντάμ του Παρισιού είχε διδακτορικό από, την, από το Πανεπιστήμιο της πόλης μου. Είναι από την ίδια πόλη. Οι αναλύσεις λοιπόν οι μακροπρόθεσμες ε, μπορούν να εντοπίσουν τέτοια στοιχεία, να απαντήσουν στα ερωτήματα τα οποία όλοι θέτουμε προφανώς. Επίση, κατά δεύτερον, απαντήσετε σε μια ερώτηση την οποία είχα, η οποία ήταν η εξή. Αν όλα τα κράτη πλήττονται, αν μάλλον συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη και όλες οι υπηρεσίες. Κάτι άλλο, μία άλλη ερώτηση. Ο, το κυβερνοέγκλημα, η κυβερνοτρομοκρατία. Ένα θέμα το οποίο τακτικά το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Η οργάνωση δηλαδή τρομοκρατικών ενεργειών μέσω του διαδικτύου ή τρομοκρατικών ενεργειών ή τα γενικά παρανομών δραστηριοτήτων εγκλημάτων. Ασχολείστε με τα θέματα αυτά και το κυβερνό έγκλημα αποτελεί ένα θέμα στο οποίο αν πρόκειται για μοναχικούς ε, λύκους, ε, ε, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν το πιστεύω αυτό απαραίτητα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ή κατά πόσον υπάρχει οργάνωση σε σχέση και με τα στοιχεία αυτά που μας παρουσιάσατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την Νάταλη. Η κυρία Κόμες έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και όλη την ε, σημαντική δουλειά που κάνει η Europol στον τομέα αυτό. Γιατί ξέρουμε πώς εξαρτώμαστε από τη συνεργασία των μυστικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών επιβολή του νόμου. Δεν μου προκαλεί έκπληξη να σα πω το γεγονό ότι βλέπω να αυξάνεται ο αριθμό των τραυματικών επιθέσεων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού. Πάντα έτσι γίνεται. Όχι στην Ευρώπη ενδεχομένω, αλλά πριν από 18 χρόνια που ζούσα στην Ινδονησία, αυτό ήταν ήδη τακτικό φαινόμενο. Και ακόμα πιο πολύ σε συνδυασμό με την απόσυρση των στρατευμάτων στη Ιράν, στη Μοσούλη, στη Συρία. Αλλά η ερώτηση που ήθελα εγώ να θέσω είναι η εξή. Καταρχά, είδαμε ότι η τρομοκρατική επιθέση στο Μάντσεστερ κάπω συνδέονταν με την Λιβύη. Όχι με τους πολίτες της Λιβύης, με πολίτες μάλλον της ε, Λιβύης που είχαν φύγει από τη Λιβύη από την οικογένεια του Καντάφη. Αλλά από ό,τι φαίνεται η Λιβύη κατέστησε καταφύγιο για πολλές τρομοκρατικές οργανώσεις. Εσείς θεωρείτε όντως ότι η Λιβύη καθίσταται πηγή και κέντρο επιμελητίας οργάνωσης, υποστήριξης. Όχι το κράτος της Λιβύης, το οποίο δεν υφίσταται. Αλλά η περιοχή, την οποία και εκμεταλλεύονται οι τρομοκρατικές οργανώσεις. Κατά δεύτερον, βρισκόμαστε τώρα με το μέσο των διαμαχών ε, Σουνιτών και Σεϊτών, με το Κατάρ επίθεση από τους Σουνίτες για την ε, συμμαχία με τον Ιράν και είδαμε και τις θερμοκρατικές επιθέσεις στο Ιράν. Πιστεύετε ότι υπάρχει σύνδεση, υπάρχει σχέση. Το στρατόπεδο των Σουνιτών προφανώς είναι το στρατόπεδο το οποίο χρηματοδοτεί και διευκολύνει την τρομοκρατία των σαλαφιστών και άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων, για να το πούμε έξω από τα δόντια. Πώς πιστεύετε λοιπόν, ε, πώς ερμηνεύετε τη σημερινή κατάσταση, αυτά που συμβαίνουν σήμερα, θα υπάρξει άλλη μια πηγή, έτσι, τρομοκρατικών επιθέσεων και άλλων τρομοκρατικών επιθέσεων. Και σε ό,τι αφορά το Μάντσεστερ στο Λονδίνο, είδαμε ότι πολλοί από αυτούς που διέπραξαν τις επιθέσεις ε, εντοπίστηκαν από το κοινό και μεταφέρθηκαν στις αρχές ε, ως ύποπτη για ριζοσπαστικές ιδέες και ενέργειες. Δεν διώχθηκαν όμως γιατί δεν υπήρχαν αρκετοί πράκτορες για την εφαρμογή του νόμου. Υπήρξε δραματική μείωση και περικοπή του προσωπικού από την κυβέρνηση των Τόρις. Πιστεύετε ότι αυτό μας ανησυχεί ιδιαίτερως, όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά παντού, γιατί αυτό αποτέλεσε μία από τη συνέπεια των προγραμμάτων λιτότητας, δραματική μείωση των πόρων και του προσωπικού στην εφαρμογή του νόμου. Όλοι, όλοι η εφαρμογή του νόμου, όλοι οι υπηρεσίες εφαρμογής του, του νόμου. Και κάτι άλλο πολύ κρίσιμο, η πρόληψη της ριζοσπαστικοποίησης. Πιστεύετε ότι οι κυβέρνησεις μας έχουν κατανοήσει ότι αυτό είναι κάτι απόλυτα απαραίτητο, γιατί δεν είναι σύμπτωση ότι πιο πολλοί από αυτούς που διαπράττουν επιθέσεις είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες και κυρίως άτομα τα οποία δεν είναι σωστά ενσωματωμένα στην ε, κοινωνία μας. Η κυρία Τσινίτη. Grazie Presidente, anch'io desidero ringraziare il direttore Navarrete per la, eh, diciamo, la, relazione che ci ha fatto sul Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους να προβλέψουμε τις τάσεις για τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Νομίζω ότι οι τάσεις τις οποίες ε, βλέπουμε με τις τελευταίες απόπειρες είναι η μη προβλεψιμότητά τους. Ε, είναι δύσκολο όταν δεν μπορούμε να προβλέψουμε λοιπόν να προλαμβάνουμε και να αντιπαρατεθούμε σε αυτές τις ενέργειες σε ορισμένες προηγούμενες περιπτώσεις υπήρχαν κάποιοι τρομοκράτες που είχαν κάνει, ε, θα έλεγα, κάποιες ενέργειες παράνομες όπως ε, στον τομέα των ποινικών. Αλλά αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών και η ανταλλαγή δεδομένων η οποία έχει υπάρξει θα πρέπει να παραλαμβάνει, να περιλαμβάνει Ε, στοιχεία τα οποία να αναφέρονται και σε αυτούς οι οποίοι έχουν βεβαρημένο παρελθόν και πιθανή επαφή με διαδικασίες βυζοσπαστικοποίησης στο εσωτερικό σαν παράδειγμα των φυλακών και στα πλαίσια των προσπαθειών απορριζοσπαστικοποίησης τι πιστεύετε ότι θα πρέπει να κάνουμε. Βλέπετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν για κοινέ πράξεις ποινικού δικαίου στη φυλακή και αρχίζουν να δρούν. Αν δεν τους παρακολουθήσουμε από την αρχή δεν μπορούμε να αποτρέψουμε ε, τις τρομοκρατικές ενέργειες τις οποίες θα προβούν. Αναφερθήκατε και στο έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Θα ήθελα εδώ να κάνω και μία άλλη ερώτηση σχετικά με τον χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στην, στον τομέα αυτό τι είδους είναι τα στοιχεία τα οποία έχετε συλλέξει, ποιες είναι οι βασικές ε, πηγές ε, χρηματοδότησης, ε, πώς γίνεται και χρησιμοποιεί η τρομοκρατία τις πιο προχωρημένες τεχνολογίες που υπάρχουν σαν παράδειγμα στη μεταφορά κεφαλαίων και άλλου είδους τεχνικά μέσα. Η τρομοκρατία έχει γίνει, θα έλεγα, όπως είπατε, απρόβλεπτη. Και γι' αυτό ακριβώς η συλλογή των πληροφοριών, η επεξεργασία των πληροφοριών και η ανταλλαγή των στοιχείων με τις επιμέρους αρχές έχει αποκτήσει πολύ μεγάλη πλέον σημασία. Χολμάια. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Ναβαρέτε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ καταρχάς για το γεγονός ότι έχετε έλθει πάλι στην Επιτροπή μας και ε, πολύ λυπάμαι που δεν ήλθα από την αρχή της παρουσίασης σας, αλλά ε, θα τα ακούσω μετά την συνεδρίαση, την πρώτη παρουσία, την, ε, το πρώτο τμήμα της παρουσίασής σας. Θα ήθελα να κάνω τρεις ερωτήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να απαντηθούν και θα ήθελα να με καθοδηγήσετε εσείς. Καταρχάς, ο, η, η λέξη κίνδυνος δεν έχει κάποιον ορισμό και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα για τα άτομα τα οποία, για παράδειγμα, ε, είναι ενδυνάμει τρομοκράτες ή επικίνδυνα. Πιστεύετε ότι στο σημείο αυτό μπορεί να υπάρξει καλύτερος ε, συντονισμό, συνεργασία και κοινό ορισμό από πλευρά των κρατών μελών, γιατί δεν μιλάμε για εκατοντάδε, μιλάμε για χιλιάδε άτομα αν ε, συνυπολογίσουμε όλο το πλαίσιο. Δεύτερον, όταν ε, ήμουν στη Γαλλία, αυτό που προσπαθήσαμε είναι να προσπαθήσουμε να έχουμε επαφή με οικογένειες, να τους δώσουμε συγκεκριμένη βοήθεια, αρρωγή, αν είναι δεθυμένοι, να δεχτούν την βοήθεια αυτή και αν είναι δεθυμένες να συνεργαστούν με τις αρχές. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια γιατί κάπως θα πρέπει να διαχωρίσουμε την ασαλαφιστική σκηνή από το σκληρό πυρήνα που πραγματικά μπορεί να, δια, να διαπράξει τρομοκρατική επίθεση. Επίσης κάτι άλλο που με σοκάρει είναι η ταχύτητα με την οποία μπορεί να γίνει η μεταστροφή ενός νέου. Δεν χρειάζονται χρόνια προετοιμασία. Φυσικά υπήρχαν ε, κάποιε κάποιες ενδείξεις και ήταν λίγο ανοιχτοί αυτοί οι άνθρωποι, αλλά... Για παράδειγμα, ένας ε, ε, νέος, ο οποίος είχε ένα φίλο, τον οποίο δολοφονήθηκε για άσχετο λόγο. Ο δολοφόνος έχει φυλακιστεί. Αλλά παρόλα αυτά, άμεσα έγινε αυτή η μεταστροφή. Θα πρέπει λοιπόν τα παιδιά Στη Γερμανία μάλλον ε, έγινε ένας έλεγχος, ε, ένα, μία μελέτη για το τι θεωρούν αρχή, ποιον θεωρούν αρχή, μεγάλη αρχή τα, οι νέοι. 86% δήλωσαν ο και όχι το κράτος. Το θέμα αυτό λοιπόν επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα του κράτους δικαίου. Δεν αναφέρθηκε καν πώς μπορούμε λοιπόν να προσεγγίσουμε τις οικογένειες αυτές ε, προκειμένου να υπάρχει δημοκρατία κράτος δικαίου και κάποιες δημοκρατικές διατάξεις στη χώρα μας. Αυτό από ό,τι φαίνεται δεν έχει περάσει ως μήνυμα. Και τέλος, ανάλυση πληροφοριών. Τώρα προέκυψε ότι υπήρξε, υπήρχαν πληροφορίες, αλλά η ανάλυση των πληροφοριών για το πόσο επικίνδυνα ήταν τα άτομα και η ανταλλαγή των δεδομένων για τα ταξίδια τους στην Ιταλία, στη Γερμανία, μέσω της Λιβύης, πάλι στην Ιταλία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ανταλλαγική ανάλυση πληροφοριών. Γιατί προκαλεί εντύπωση το γεγονός όταν ξαφνικά ένα αλαφιστή ταξιδεύει στη Λιβύη ακόμα και αν έχει οικογένεια εκεί. Δεν είναι και φέρετρο η Λιβύη. Είναι χώρος ρίζος παστικοποίησης και υψηλής εγκληματικότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε τις ερωτήσεις μου. Ο Πρόεδρος, όπως βλέπετε, οι συναδελφοί γνωρίζουν αυτό το θέμα εις βάθος και θέτουν τις ερωτήσεις αυτές και νομίζω ότι όλα αυτά χρήζουν εμβελεχούς μελέτης στο θέμα της ριζοσπαστικοποίησης θα είναι δύσκολο να τα συνενώσετε όλα αυτά τα θέματα και να ανταποκριθείτε αν θέλετε στο ύψος των ερωτήσεων. Πείτε μας όμως η Γιουροπόλ, σε τι φάση είναι, τι διαπιστώνει στην παρούσα φάση, αν μπορείτε. Um, το ξέρω ότι είναι μεγάλο το καθήκον αυτό και είναι μεγάλες ερωτήσεις που σας έθεσαν οι πέντε συνάδελφοι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Μερικές φορές θέτω και εγώ τα ίδια ερωτήματα. Προσπαθώ να αναλύσω τα δεδομένα, κάνω υποθέσεις και προσπαθώ να κάνω και κάποιες προβλέψεις έτσι ώστε να προλαμβάνονται τέτοιου είδους δράσεις όσο μπορεί κανείς περισσότερο. Τώρα μου ζητάτε να προσπεράσω και τα όρια τη ΤΙΣΑ και ε, θα προσπαθήσω να το κάνω και να αξιολογήσω το πώς βρισκόμαστε σήμερα και το αν μπορούμε να κάνουμε καλύτερο και περισσότερο ε, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε. Εγώ σας παρουσίασα την εικόνα για το 2016. Γνωρίζετε τα θέματα αυτά της ερωτήσεις σας. Βλέπετε πόσο ρευστή και ε, σε συνεχή αλλαγή είναι η κατάσταση που περιβάλλει την τρομοκρατία. Πρέπει και εμείς λοιπόν να είμαστε ευέλικτοι, ευκίνητοι και ευπροσάρμοστοι όπως είναι οι τρομοκράτες. Υπάρχουν δύο βασικά θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να ατύχουν βελτιώσεων. Καταρχάς, ανταλλαγή πληροφοριών. Έχει υπάρξει λοιπόν προσπάθεια ποσοτική αλλά και ποιοτική πρέπει να υπάρξει, όχι μόνο σε επίπεδο Europol, εμείς είμαστε μια πλατφόρμα. Απλά διευκολύνουμε την ανταλλαγή. Η πραγματική ανταλλαγή γίνεται σε διμερές επίπεδο και νομίζω ότι δουλεύει καλά. Η διμερή συνεργασία βέβαια ε, συνήθως δεν αφήνει ίχνη. Ενώ μια πολυεθνική πλατφόρμα έχει μνήμη και ε, καταγράφει όλα τα στοιχεία αυτά. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορά μεγάλη από ό,τι νομίζω ανάμεσα στη διμερή συνεργασία και τη συλλογική πλατφόρμα. Μπορούμε όμως να συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον. Έχει υπάρξει λοιπόν ισχυρή εξέλιξη στις διμερείς σχέσεις. Θα πρέπει επίσης δύο παράγοντες να λάβουμε υπόψη μας και να δούμε τι ακριβώς είναι σημαντικό. Πρώτον, η ταχύτητα. Σε άλλους τομείς μπορούμε να είμαστε πιο αργοί, αλλά τώρα πρέπει να είμαστε ταχύτατοι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ε, κάτι να εξελιχθεί από μόνο του θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δράσουμε γρήγορα και θα πρέπει να είμαστε ακριβείς στις πληροφορίες, στις τεχνικές που δίδουμε. Δεν πρέπει να υπάρχουν λάθη. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την ανάληψη δράσης, αλλά πρέπει να είμαστε επακριβείς στα στοιχεία. Τώρα για τις τάσεις. Νομίζω ότι το βασικό κομμάτι της αστυνομικής δουλειάς ε, είναι να ε, βρει κάποιους συγκεκριμένους δρόμους ε, και μορφές που θα μας επιτρέψουν να προλάβουμε τις τρομοκρατικές ενέργειες. Οι τρομοκράτες έχουν γίνει όμως όπως είπα απρόβλεπτοι και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουν γίνει και μία αποτρέψιμη. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν μέσω των αναλυτικών εκθέσεων της συλλογή πληροφοριών και της συγκράτησης της μνήμης των στοιχείων αυτών είναι να εντοπίζουμε σωστά τους ύποπτους για τρομοκρατία, να βλέπουμε τι κινδύνους δημιουργούν στην παγκόσμια ασφάλεια και στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και να αναλαμβάνουμε δράσεις έτσι ώστε οι πιθανοί τρομοκράτες να ριζοσπαστικοποιούνται και να προβαίνουν στις ε, πράξεις αυτές. Αυτός είναι ο στόχος, να προσπαθήσουμε να τους καταστήσουμε προβλέψιμους και τότε θα μπορούμε να τους καταστήσουμε και αποτρέψιμους. Στην ουσία λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε τώρα είναι κάποιες ε, εκθέσεις αναλυτικές σε κάποια φαινόμενα μακροπρόθεμα όπως σαν παράδειγμα ποια είναι τα κίνητρά τους, γιατί κάνουν τις συγκεκριμένες επιλογές, γιατί ακολουθούν τις συγκεκριμένες διαδρομές, ποιες μπορεί να είναι οι διαδικασίες έβρεσης των στόχων τους στο μέλλον, τι μπορεί να βοηθήσει ε, τον αξιωματικό της ε, ε, υπηρεσίας ασφαλείας στην πρώτη γραμμή να αντιμετωπίσει τις συνθήκες που θα του δώσουν το ποιος είναι πιθανός τρομοκράτης και να δούμε πώς μπορούμε να αποτρέψουμε επιθέσεις σε στρατιωτικές και αστυνομικές μονάδες, γιατί και αυτό είναι μία τάση. Αυτές είναι οι πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσουμε με τα κράτη-μέλη στο μέλλον σχετικά με τον κυβερνοχώρο. Εδώ δεν έχουμε ενδείξεις ότι οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν κάποια μέσα στο διαδίκτυο ε, για να πετύχουν τον στόχο τους. Αν το κάνουν θα τους παρακολουθήσουμε, μέχρι τώρα όμως έχουν προθέσεις να το κάνουν, αλλά προς το παρόν δεν έχουν τις ικανότητες και τα μέσα να δημιουργήσουν προβλήματα ξεπερνώντας ε, τα εμπόδια τα οποία βάζουμε εμείς και τα συστήματα προστασίας ε, των δικτύων μας. Ε, υπάρχει όμως το θέμα της προπαγάνδας, εμείς θα πρέπει να υπογραμμίζουμε το ποια είναι αυτή η προπαγάνδα, να την εντοπίζουμε και να μετριάζουμε τις συνέπειες της προπαγάνδας αυτής έτσι ώστε να μην μπορεί ο κόσμος να ε, ριζοσπαστικοποιείται και θα πρέπει να ελέγξουμε καλύτερα και το λεγόμενο dark web, το σκοτεινό διαδίκτυο, ε, γιατί το χρησιμοποιούν για αγορά όπλων, για προσπορισμό εσόδων, ε, όχι μόνο στην τρομοκρατία, αλλά ευρύτερα στην εγκληματική δραστηριότητα. Δεν θα πρέπει να υπάρξει όμως χώρος προστασίας, δεν θα πρέπει να υπάρξει ασφαλές καταφύγιο. Ε, χρησιμοποιούν πολλά μέσα βέβαια, όπως επίσης και εναλλακτικά νομίσματα όπως το bitcoin. Ε, η τρομοκρατική δραστηριότητα ε, μέχρι τώρα είναι ευθυνή. Αυτό που είναι ακριβό είναι η χρηματοδότηση. Αν είσαι μόνος σου δεν χρειάζεσαι πολλά. Παίρνεις ένα αυτοκίνητο, νοικιάζεις ένα αυτοκίνητο και κάνεις αλλά υπάρχει οργανωμένος τρόπος τρομοκρατικής ε, ομάδας, κάτι το οποίο έχει οικονομικές ε, συνέπειες, κοστίζει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι είναι οι νέες τεχνολογίες τις οποίες έχουμε για το Μάντσεστα. Ξέρετε ότι η έρευνα γίνεται από τις αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες συλλογής πληροφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές. Είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς την κατάσταση όπως έχει. Αλλά τα προφίλ των δραστών είναι παρόμοια με αντίστοιχα που έχουμε ζήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ίσως να μην αναφέρθηκα στο ότι υποστηρίζουμε, παρακολουθούμε 100 127 times. 127 περιπτώσεις. We were supporting one or two member states οι περιπτώσεις αυτές μερικές φορές δεν συνδέεται μεταξύ, δεν συνδέονται μεταξύ τους. Ας πούμε το Μάντσεστερ δεν συνδέεται με το Λονδίνο ε, και αντίστοιχα κάποιες άλλες δράσεις και παρεμβάσεις μεταξύ τους δεν συνδέονται. Δεν είναι ένα δίκτυο δεδομένο δηλαδή και αυτό είναι καλό. Από την άλλη βέβαια όσο δεν είναι δικτυωμένοι τόσο δύσκολο είναι να προλαμβάνει κανείς τις ενέργειες αυτές. Όταν κάποιος λειτουργεί μόνος του λοιπόν, με μονομένα, ε, είναι δύσκολο να ε, εντοπιστεί. Είναι πιο δύσκολο και για τις αστυνομικές υπηρεσίες να συλλέξουν πληροφορίες, να φτιάξουν ένα σωστό προφίλ και να αναλάβουν δράση. Γιατί η αξιολόγηση των κινδύνων έχει προτεραιότητες. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω από κάθε ύποπτο, δεν μπορούμε να παρακολουθούμε όλους τους υπόπτους 24 ώρες το 24ωρο. Do better. So it's about risk assessment and prioritization. And we need all the information that we have on this one. Τώρα τα κράτη-μέλη πρέπει να υποστηρίξουν την Europol για να μπορέσουμε και εμείς να αποδώσουμε καλύτερα. Τώρα για την ε, σύγκρουση Σία και Σούνη. Αυτό θα επηρεάσει λίγο τα θέματα ασφαλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ε, βίαιες δυνάμεις και στις δύο πλευρές που έχουν επιτεθεί η μία στην άλλη. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους Σιωσίτες, ούτε για τους Σουνίτες, ούτε για τους Χριστιανούς, Μουσουλμάνους κτλ. Η σύγκρουση αυτή είναι κάτι το οποίο θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα δυστυχώς. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Να αναφερθώ σε σχέση με το ότι η θρησκευτική τρομοκρατία δεν είναι ο μοναδικός λόγος για να γίνει κανείς τρομοκράτης. Ε, υπάρχουν θέματα ανταπόδοσης, υπάρχουν θέματα ακυρεοφρονισμού υπάρχουν γενικά πάρα πολλές εξηγήσεις και δικαιολογίες και προσωπικοί λόγοι και πολλές φορές οι δολοφονίες γίνονται ακριβώς μετά από ριζοσπαστικοποίηση και αυτή θα πρέπει να αποτρέψουμε. Εδώ είναι σημαντικός ο ρόλος των κοινωνικών επιστημόνων, των κοινωνικών οργάνων, των ψυχολόγων του κοινού και των κοινωνικών δικτύων. Δεν έχουμε εναλλακτικό δρόμο, δεν έχουμε μια διαφορετική ρητορική, δεν μπορεί η αστυνομία να το κάνει αυτό, το κοινοβούλιο μπορεί να το κάνει, το κοινό μπορεί να το κάνει, οι δημοσιογράφοι μπορούν να το κάνουμε, μπορούν να λέμε στους ανθρώπους αυτούς ότι δεν κάνουν σωστά και έτσι ε, θα πρέπει να στέλνονται στη φυλακή αυτή η δουλειά της αστυνομίας όταν κάποιοι παραβιάζουν τον νόμο. Αλλά σε επίπεδο κοινωνικών μέσων δικτύωσης και στον τομέα των εκπαιδευτικό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα Νομίζω λοιπόν ότι όντως υπάρχει καλύτερη συνεργασία, αλλά όπως είπε και η κυρία Χολμάγερ, ε, ακόμα υπάρχουν κενά. Χρειαζόμαστε όλο και περισσότερες πληροφορίες, γιατί κάθε περίπτωση διαφέρει από την προηγούμενη. Και επομένως ε, δεν αρκεί να πούμε ότι το Βερολίνο διαφέρει από το Μάντσεστερ, το Παρίσι διαφέρει από το Βέλγιο, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Όχι, το αντίθετο. Μπορούμε. Προσπαθούμε να ταυτοποιήσουμε κάθε και να περιγράψουμε κάθε μία περίπτωση, κάθε μία ξεχωριστή περίπτωση και να πάρουμε στοιχεία τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε άλλες περιπτώσεις. Μετά τις επιθέσεις στο Μάντσεστερ, στο Λονδίνο, αλλά και μετά από το Παρίσι κλπ. Το πιο σημαντικό ερώτημα που πρέπει να ε, θέσουν τα κράτη-μέλη είναι τι, τι, συμβαίνει, ε, τι συνέβη, πόσα είναι τα θύματα κτλ. Και το δεύτερο είναι ποιος το έκανε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Τι συνέβη και ποιος το έκανε. Και για την ασφάλεια των υπολείπων χωρών, πίσω από το ποιος είναι ο υπεύθυνος, το κύριο ερώτημα είναι πώς, πώς συνέβη αυτό και γιατί συνέβη αυτό το κράτος μέλος που το αφορά που έχει δεχτεί την επίθεση πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα του τι συνέβη ακριβώς και πώς θα το ξεπεράσει και ε, οι, άλλοι, ε, οι άλλες χώρες θα πρέπει να ε, αναρωτηθούν πώς μπορούν να αποφευχθούν τέτοιου είδους περιστατικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μανουέλ Ναβαρέτε. Πραγματικά σας ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτό το απόσταγμα σοφίας το οποίο μας δώσατε βάσει τις εμπειρίες σας και τις εμπειρίες ε, των συναδέλφων σας ε. Αναμφίβολα, πολλή συνεργασία θα ε, υπάρξει, πολλή δουλειά θα κάνουμε όσον αφορά την αντιτομοκρατία. Επίσης θα συζητήσουμε και το αντιτρομοκρατικό αφήγημα των μέσων ενημέρωσης. Εδώ υπάρχουν ε, κάποια κενά τα οποία πρέπει να καλυφθούν, αλλά και αυτή η σύντομη αλλά υψηλής ποιότητα συζήτηση ήταν πάρα πολύ ε, σημαντική. Είναι κρίμα που ήταν πέμπτη απόγευμα, αλλά σας ευχαριστούμε που ήρθατε ε, για να μοιραστείτε μαζί μας την εμπειρία σας. Έχουμε πολλούς επισκέπτες ε, που ήρθαν στη διάρκεια της συζήτησης, την οποία ελπίζω ότι θα έχουν βρει ε, ε, ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για κάποια αντιπροσωπεία επισκεπτών της κυρία Πίσμπακ. Σας καλωσορίζουμε όλους λοιπόν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Και νομίζω ότι ε, συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις χειροκροτούμε. Γιατί να μην το κάνουμε και αυτή τη φορά. Ακόμα και τους, δικαστη... τους δικηγόρους τους, ε, ε, τους ε, χειροκροτούμε. Ελπίζω ότι καταλάβατε όλοι το χιούμορ μου, γιατί καμιά φορά τον περνάει από μετάφραση χαλάει λίγο. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και τα, ε, τους βουλευτές που ήρθαν και συμμετείχαν σε αυτή την συζήτηση. So, colleagues, we go to the final point of... Τελευταίο σημείο της μερισσία διατάξεως, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε το σημείο 17, μόλις ολοκληρώσουμε το 16. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους αδέλφους που είναι εδώ, τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Η ανακοίνωση αφορά την προστασία των παιδιών μεταναστών. Είχαμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη, υπάρχουν και άλλες ταυτόχρονες συνεδριάσεις. Ε, δεν είναι τυραμόλες τα μέλη, δεν μπορούν να είναι παντού. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πριν από λίγο καιρό η Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, ε, δημοσιοποίησε την ανακοίνωσή της σχετικά με την προστασία των παιδιών μεταναστών. Δεν χρειάζεται ε, να σας πω ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ ε, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ε, κυρίως αυτοί που δεν έχουν καμία μορφή συνοδείας ή προστασίας και επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν τέτοιες προτάσεις στα πλαίσια του κοινού προγράμματος ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, φέτος ε, θα αρχίσει να λειτουργεί ένα ευρωπαϊκό ε, δίκτυο επιμελητίας ακριβώς για αυτούς τους ασυνόδευτους ανήλικους. Θα δώσω το λόγο στον Στίβεν Ράιαν από την DG Home και την Κάρα Δάμο από την DG Δικαιοσύνης Justice για να μας παρουσιάσει αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Θα ξεκινήσουμε με τον Στίβεν, όχι, Ξέρω ότι ο συνάδελφος έδειξε την Κιάρα, αλλά νομίζω θα ξεκινήσουμε από τον Στίβεν. Όχι, από την Κιάρα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για να παρουσιάσουμε την ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χρειαζόμαστε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προκειμένου να παραμείνουν στο κέντρο τη πολιτική ατζέντα τα συμφέροντα και τα το θέμα των προστασίας των παιδιών και να σας ε, πω γιατί εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ανακοίνωση αυτή το 2015 και 2016 30% των ετούντων άσυλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν παιδιά και αυξάνεται το ποσοστό παιδιών που ετούνται άσυλο τα τελευταία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 350.000 παιδιά έφτασαν μέσα από τη θάλασσα το 2015 στην Ευρώπη. Φυσικά αυτό κάνει τη διαχείριση των ζητημάτων αυτών στα κράτη-μέλη πιο δύσκολη και ουσιαστικά επιδεινώνει προβλήματα τα οποία ίδια, ήδη υπήρχαν σε ό,τι αφορά τα παιδιά μετανάστες. Τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο έτος ε, έγιναν διάφορες συζητήσεις ε, για με ακτιβιστέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα θέματα αυτά και επίσης ακούσαμε πολλές μαρτυρίες από τα ίδια τα παιδιά. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πολύ δύσκολη. Απαράδεκτη, μάλιστα, από κάποιες απόψεις. Και έτσι εκτιμούμε την ε, υποστήριξη και όλη τη δουλειά του, της ε, ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δικαιώματα των παιδιών. Οι βουλευτές της οποίας έχουν παίξει πάρα πολύ σημαντικό και επικοδομητικό ρόλο στις διαβουλεύσεις. Τον Νοέμβριο του περσινού έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εστιάστηκε στα θέματα των δικαιωμάτων των παιδιών μεταναστών και εντοπίζοντα τέτοιες ανάγκες ε, καταλήξαμε στις ε, πιο κατεπίγουσες δράσεις οι οποίες χρειάζονται να αναλευθούν. Στην ανακοίνωση αυτή λοιπόν, ε, καταρχάς αναφέρουμε ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες των κρατών μελών προκειμένου να ανέλθουν στο ύψος των περιστάσεων και θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να κάνουν τα απαραίτητα για την προστασία των παιδιών και επίσης ε, να βοηθήσουμε τα παιδιά να ζητούν, να γνωρίζουν και να ζητούν την εφαρμογή των δικαιωμάτων τους. Φυσικά πρώτο συμφέρον, πρώτο μέλημα είναι τα δικαιώματα των παιδιών και η προστασία των παιδιών και όπως σας είπα η ανακοίνωση εστιάζεται στα πιο κρίσιμα πραχυπρόθεσμα ζητήματα η... το φαινόμενο των παιδιών μεταναστών περιλαμβάνει πολλά παραπάνω πέρα από τους ασυνοδευτούς ενηλίκους όπως για παράδειγμα την επανένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους και Θέλουμε να αναπτύξουμε λοιπόν το δυναμικό και τα συστήματα προστασίας των παιδιών. Αυτό σε μέσο και μακρό πρόθεσμο επίπεδο στα εθνικά μας συστήματα. Θα ήθελα να αναφέρω δύο ζητήματα πρωτού δώσω το λόγο στον συνάδελφο από τη Γενική Διεύθυνση Home. Καταρχάς, η αποτελεσματική και η Τα παιδιά μετανάστες όχι μόνο χρειάζονται προστασία. Χρειάζεται και σταθερότητα, συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν μόνο σε προασπίζονται τα δικαιώματά του με τον καλύτερο τρόπο, θεωρούμε. Και αυτό δεν σχετίζεται μόνο με τη διαδικασία αίτηση ασύλου, παρά το γεγονό ότι τώρα σε αυτό επικεντρωνόμαστε. Αυτό αποτελεί κεντρικό στοιχείο σε ό,τι αφορά τα παιδιά μετανάστες, αλλά φυσικά περιλαμβάνεται και το θέμα της σωστής πρόσβαση στις διαδικασίες ε, λήψης απόφασης, ε, επαφή με τις οικογένειες και το καθεξής. Και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το διασυνοριακό στοιχείο εδώ. Σε ό,τι αφορά τους ε, κυδεμόνες, ζητούμε λοιπόν από τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις ιδιώδους συνεργασίες όπως αυτή που Προβλέποντα στις Βρυξέλλες 2. Στη συμφωνία αυτή, μία από τις δράσεις λοιπόν, που ανακοινώσαμε είναι η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου για την κυδαιμονία. Αρχίσαμε να εργαζόμαστε από αυτού και θα συνδεθούμε με την, ε, με την ομάδα εμπειρογνωμών την άλλη εβδομάδα στις 16 Ιουνίου. Σκοπός είναι να υπάρξει χρηματοδότηση της ε, Ένωσης για την πρωτοβουλία αυτή και σε ό,τι αφορά την υποδοχή θα πρέπει να υπάρχει ε, να υπάρχουν ε, αναδόχες οικογένειες οι οποίες θα βασίζονται πιο πολύ στον πυρήνα της οικογένειας και επίσης ε, θα πρέπει να εξετάσουμε την διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα σε, στη λύση της αντικειτικής κράτησης των παιδιών. Αυτό πραγματικά αποτελεί κατεπίγουσα ανάγκη. 6 και 7 Νοεμβρίου θα γίνει μια διάσκεψη για το θέμα αυτό της κράτησης των παιδιών και την προώθηση των εναλλακτικών από πλευρά των κρατών μελών προς τη λύση αυτή. Ελπίζω λοιπόν το κοινοβούλιο αυτό και οι βουλευτές θα συμμετάσχουν. Σήμερα συζητάμε στο Συμβούλιο των Υπουργών ε, ένα κοινό συμβούλιο εγκρίνει, ελπίζω εγκρίνει τις βάσεις για την ανακοίνωση αυτή και καλεί τα κράτη-μέλη να εφαρμόσει και να αναλάβει δράση και να εφαρμόσει μέτρα για να υλοποιηθούν οι στόχοι της ανακοίνωσης. Το οποίο θεωρούμε ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα πρόοδου γιατί οι πιο πολλές ε, ενέργειες εξακολουθούν να εξαρτώνται από την πολιτική βούληση των χωρών που συμμετέχουν στο Συμβούλιο. Αυτά και θα δώσω το λόγο στο Στίβεν Ράιεν από την Γενική Διεύθυνση Home για τις άλλες δράσεις. Ευχαριστώ, κιέρα. Ευχαριστώ και σας, κύριε Πρόεδρε. Να συμπληρώσω την παρουσίαση του συναδέλφου, τη συναδέλφου, δίδοντας κάποιες λεπτομέρειες για τις συγκεκριμένες δράσεις, τις οποίες έχει παρουσιάσει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της. Υπάρχουν κάποιες κατεπίγουσες δράσεις, οι οποίες θα πρέπει να αναλυφθούν τάχιστα, για την ενίσχυση της διαμεσοριακής συνεργασίας έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εθνικό επίπεδο και τοπικό επίπεδο να συμμετέχουν. Να υπογραμμίσω ορισμένες από τις βασικές δράσεις που πρέπει να αναλυφθούν για να βελτιώσουν τη θέση των παιδιών μεταναστών με σωστό τρόπο. Θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι τα παιδιά θα καταγράφονται άμεσα αυτή τη στιγμή φτάσουν σε κοινοτικό έδαφος και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα αμέσως έτσι ώστε να μην κηρύσσονται αγνοούμενοι. Διατρέχουν ειδικού κινδύνους εκμετάλλευση σωματεμπορίας και όπως γνωρίζετε ο αριθμός των παιδιών τα οποία δηλώνονται ότι αυτή τη στιγμή ε, είναι, έχουν απολεστεί είναι αγνοούμενα, είναι υψηλότατος. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να συλλέγουν συγκρίσιμα στοιχεία και να διευκολύνουν την παρακολούθηση και εντοπισμό των αγνοούμενων παιδιών και των οικογενειακών του συνδέσμων. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα απαραίτητα πρωτόκολλα έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των παιδιών αυτών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πάρα πολλές ευθύνες σε σχέση με την διαδικασία ε, εντοπισμού και καταγραφής και με συγκεκριμένο τρόπο ζητάμε εμείς να υπάρξουν ειδικοί οι υπάλληλοι που ανασχολούνται με το θέμα αυτό για την καταγραφή τους, να γίνεται αξιολόγηση των μεμονωμένων περιπτώσεων της ηλικία των παιδιών με μεθόδους μη παρεμβατικές, χρησιμοποιώντας ένα διεπιστημονικό τρόπο που να περιλαμβάνει και ψυχολογικές τεχνικές και γι' αυτό οι διάφορες ε, υπηρεσίες ασύλου ε, προσπαθούν να βρουν τις σωστές μεθόδους για την αξιολόγηση της ηλικία. Απαιτείται επίσης ένα αναθεωρημένο σύστημα το οποίο να προστατεύει καλύτερα από ό,τι σήμερα τα παιδιά που έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία τη στιγμή που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να προστατευθούν τα συμφέροντα των παιδιών στο σύνολο των νομικών μέσων τα οποία έχουμε θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι οι ανήλικοι εντοπίζονται γρήγορα οι εκπρόσωποι που θα αναλάβουν την κυδαιμονία τους να το κάνουν αυτό και να βρίσκονται με υψηλή επίσης ταχύτητα και να υπάρχουν αποδεκτές συνθήκες υποδοχής για τα παιδιά αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά από τους δύο συνομοθέτες, το Συμβούλιο δηλαδή και το Κοινοβούλιο, να καταλήξουν σε μια συμφωνία σε αυτά τα τμήματα του πακέτου. Παράλληλα ζητάμε από τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν τις αιτήσει που καταφέτουν τα παιδιά για άσυλο κατά προτεραιότητα. Ζητάμε από τα κράτη-μέλη, όπως ακριβώς το έχουμε κάνει επανειλημμένα στο παρελθόν, να δώσουν προτεραιότητα στα θέματα της επανεγκατάστασης των παιδιών από την Ιταλία και την Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά για αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης, και αυτό έχει σημασία, ότι είναι σημαντικό να βρεθεί μια διαρκής λύση προς όφελος, των παιδιών αυτών. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ενταχθούν ενταχθούν ε, καλύτερα στην ε, ε, στα, στις νέες τους χώρες και βεβαίως θα πρέπει ε, με κάθε τρόπο να προωθηθεί η οικογενειακή επανένωση. Ε, θέλουμε παιδιά καλά ενσωματωμένα που θα γίνουν μέρη ε, άρρηκτα της κοινωνίας μας. Θέλουμε επομένως πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην, στις υπηρεσίες υγείας, εκμάθηση της γλώσσας της χώρας και κτλ. Ε, ε, ε, Βεβαίω έχουμε και κάποια πολύ καλά παραδείγματα, πρόσβαση σε στέγαση και εκπαίδευση και τα και αυτό θα πρέπει να γίνεται με τρόπο συμπεριληπτικό και τρόπο που δεν θα οδηγεί σε ξενοφοβία και ρατσισμό. Η ανείχνευση των οικογενειών και η βελτιστοποίηση των ε, μέτρων ένταξης στη χώρα υποδοχής είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όλα αυτά ε, τα υπογραμμίζουν τα κράτη-μέλη και τα υποστηρίζουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση χρηματοδοτεί οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και άλλες οργανώσεις οι οποίες δουλεύουν στη βάση με τέτοια προγράμματα. Το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω σχετίζεται με την αντιμετώπιση των αιτίων που οδηγεί, σε αυτά, οδηγεί αυτά τα παιδιά στο να ε, πάρουν ε, το δύσκολο δρόμο και να ακολουθήσουν ε, αυτήν την επικίνδυνη οδό. Ο πόλεμος και η φτώχεια είναι κάποια από τα αίτια αλλά βεβαίως ε, θα πρέπει να καλύψουμε και τις ελλείψεις όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Ε, η κατάσταση των παιδιών σε πολλά μέρη του κόσμου, ε, συμπεριλαμβανομένων και των χωρών από τις οποίες περνούν οι διαδρομές μεταναστευτικές, πραγματικά είναι κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές και επομένως καλή, καλή και καλύτερη συνεργασία μεταξύ και των τρίτων χωρών όσον αφορά την προστασία των παιδιών. Επίσης, ε, πρέπει να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με εκπροσώπους ε, της ε, κοινωνίας των πολιτών και με μη κυβερνητικέ οργανώσεις στις χώρες αυτές. Δυστυχώς πρέπει να σας διακόψω γιατί θα φύγουν οι βουλευτές. Ναι, ναι, τελειώνω, τελειώνω. Επομένως θα πρέπει με τις χώρες προέλευσης ε, να ξεκινήσουμε ιδιαίτερη συνεργασία ε, και βεβαίως να βρούμε τρόπους ε, να διώξουμε από την εικόνα τις εγκληματικέ οργανώσεις και τις συμμορίες. Επίσης θα πρέπει να ενδυναμώσουμε το πρόγραμμα επανεγκατάστασης κυρίως για τα παιδιά, για τους ανήλικους αυτούς που δεν μπορούν μόνοι του να συνεχίσουν το δρόμο έτσι ώστε να βρούνε ασφαλές καταφύγιο σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ. Ε, ξέρετε, έχουν ε, οι βουλευτέ μας ε, ε, πτήσεις που πρέπει να πάρουν. Και δυστυχώς πρέπει να φύγουν λοιπόν αυτό, γι' αυτό σα διέκοψα. Σχετικά με την ανακοίνωση αυτή, πραγματικά είναι κρίσιμη σημασίας. η Άννα Γκόμες και η κυρία Κιανίτσι ε, όσοι πήγαν και στην Ελλάδα και έκαναν μια σχετική αποστολή ζητούν σωστή επιμελητία, ζητούν κυδεμόνευση των παιδιών αυτών. Αυτή είναι η απόλυτα πρώτη προτεραιότητα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί διαβάζοντας αυτή την ανακοίνωση γιατί ε, η ενσωμάτωση εξαρτάται από το κόστος που θα ε, παρουσιάσει η ε, ενσωμάτωση αυτή στους προϋπολογισμούς της κοινωνικής ασφάλισης και τους λοιπούς προϋπολογισμούς των χωρών. Δεν είναι εύκολες λύσεις αυτές. Ε, και ξέρετε ότι τα συστήματα προστασίας των παιδιών διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Επομένως, ε, ε, εδώ είναι πραγματικά μεγάλη η πρόκληση. Εξαιρετική, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ανακοίνωση. Τώρα βέβαια πρέπει να υλοποιηθεί. Ήψη τη σημασία λοιπόν, το ξαναλέω, είναι αυτή η ανακοίνωση και μα ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα προσπαθήσουμε όλοι να ε, βάλουμε αέρα στα πανιά της έτσι ώστε να προχωρήσει. Ε, και πραγματικά σας ευχαριστούμε ε, που μας είπατε, μας, μας παρουσιάσατε την ανακοίνωση αυτή. Η Κατερίνα Ανίτσι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους της Κομισιόν όχι μόνο για την ε, ε, καλή παρουσίαση του περιεχομένου ε, της ανακοίνωσης, αλλά και γιατί ε, είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με τη συνάδελφο Κοράτσα Μπίλτ στα πλαίσια της ε, δικής της ε, εργασίας. Θα ήθελα επομένως να ευχαριστήσω και για την εργασία που έγινε στα πλαίσια του Intergroup. Όσον αφορά την, το συγκεκριμένο κείμενο, την ανακοίνωση για την προστασία των παιδιών μεταναστών, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι πολύ δυστυχώ οι ανήλικοι οι οποίοι ξεκινούν δραματικά ταξίδια ε, και το, η ανακοίνωση περιλαμβάνει πάρα πολλά ενδιαφέροντα ε, και σημαντικά στοιχεία. Όπως είπες και εσύ, ε, το θέμα της, επιμελίας, της, συγγνώμη, της επιμέλειας, το θέμα του δικτύου κυδαιμονίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αφορά όλους τους ανήλικους. Θα πρέπει οπωσδήποτε οι κυδαιμόνες αυτοί να είναι προετοιμασμένοι καλά. Ε, γιατί πρέπει από την ώρα που φτάνει ο ανήλικος στο hot spot να πέσει σε καλά χέρια για να, μπορέσει, ε, να μπορέσουν οι υπεύθυνοι με τα λόγου γνώσεως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των παιδιών αυτών. Ένα άλλο σημείο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς το έχουμε πει επανειλημμένα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αλλά και στο Intergroup δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιαδήποτε μορφή κράτησης ε, για τους ε, ε, ανήλικους μετανάστες. Αυτή πρέπει να είναι μια δέσμευση ισχυρότατη και της Κομισιόν και όλων των χωρών και θα πρέπει να βρεθούν εναλλακτικέ λύσεις και επομένως χαίρομαι γιατί αναφέρθηκε και σήμερα ε, το, ε, η θέσπιση της ε, οικογενειακής εστίας γιατί οι νέοι, αυτά τα παιδιά τα οποία ξεφεύγουν από τραυματικές καταστάσεις θα πρέπει να, μπορεί, να μπορούν εύκολα να ενταχθούν στη νέα κοινωνία, στη χώρα υποδοχής. Και ε, θα πρέπει επομένως να καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις επιμέλειας, κυδαιμονίας, ε, ε, εκπαίδευσης κλπ. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά άλλα στοιχεία πολύ σημαντικά που αφορούν την άφηξη και την υποδοχή και την ενσωμάτωση. Αλλά το πιο σημαντικό είναι όλοι όσοι θα έρθουν σε επαφή με τον ανήλικα, να, ανήλικο να είναι σε θέση να τον κατανοήσουν και να τον βοηθήσουν. Αυτό που υπογράμμισες και εσύ είναι πάρα πολύ σωστό ε, και βεβαίως χρειάζεται, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, οικονομική στήριξη, γιατί δεν χρειάζεται μόνο υποδοχή. Ε, ο, ο ανήλικος χρειάζεται και ε, υποστήριξη και η υποστήριξη κοστίζει. Η χώρα μου την δίνει την υποστήριξη αυτή, αλλά νομίζω ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να δεσμευτούν και επομένως και να βάλουν και το χέρι στα τσέπη. Ε, τώρα, η, τα στοιχεία τα οποία μας δίνει η ανακοίνωση της Κομισιόν θα πρέπει πλέον να μεταφραστούν ε, σε συγκεκριμένες, ε, σε συγκεκριμένες ε, δεσμεύσεις και σε συγκεκριμένα ε, μέτρα. Θα πρέπει όλες ε, οι χώρες να ακολουθήσουν και να υλοποιήσουν τα στοιχεία αυτά. Οπουδήποτε βρίσκονται παιδιά τα οποία είναι τα πιο απροστάτευτα θύματα των καταστάσεων. Δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις περιπτώσεις να μην δείξουμε αλληλεγγύη και ακόμα περισσότερο δεν είναι δυνατόν να μην δείξουμε την υπευθυνότητα ε, που πρέπει να έχουμε. Ε, έχουμε ευθύνη για τα παιδιά αυτά, εμείς όλοι. Και γι' αυτό ευχαριστώ την Κομισιόν για αυτή την πάρα πολύ σημαντική εργασία ε, και καλό όλους μας, τον καθένα στην χώρα του, να βοηθήσει έτσι ώστε να αναλυφθούν οι απαραίτητες υποχρεώσεις. Εξαιρετικά τα είπες, Κατερίνα. Άννα. Και εγώ ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δουλειά αυτή και θα ήθελα πραγματικά να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει πιο πολύ. Και παραπάνω δουλειά. Να είναι πολύ δυναμικό το πολιτικό μήνυμα το οποίο θα στέλνουν στα κρατημέλη και να μην μπορούν να συνεχίσουν να το αγνοούν. Γιατί μιλάμε για την προστασία των πλέον ευάλωτων. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο σοκαρισμένοι ήμασταν όταν η αστυνομία στο Μάλμο μας είπε ταραγμένοι πως τους είχαν αφαιρέσει κονδύλια τα οποία χρησιμοποιούνταν για να ψάξουν να βρουν αγνοούμενα παιδάκια, ε, μετανάστες. Αν, αν ήταν αυτά τα παιδιά α, σουηδάκια, θα είχαν πολύ παραπάνω πόρους. Είναι και το θέμα της ασφάλειας, γιατί προφανώς αν τα παιδιά αυτά αγνοούνται, θα τα εκμεταλλευτούν τα εγκληματικά δίκτυα. Αυτό είναι θέμα ασφάλειας λοιπόν και θα πρέπει να το καταλάβουν τα κράτη-μέλη. Δεν βλέπω να κάνει σκληρές συζητήσει και διαπραγματεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα κράτη-μέλη. Είναι εξωφρενικό το ότι η επανένωση των οικογενειών δεν χρησιμοποιείται σε ό,τι αφορά τα παιδιά μετανάστες. Αυτά τα παιδιά είναι πρόσφυγες, έχουν επιβιώσει από φρικτές συνθήκες, έχουν γίνει πρόσφυγες, ακόμα και αρχικά ήταν μετανάστες. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, το βασικό ζήτημα είναι να εστιαστούμε στα παιδιά, τα παιδιά στην Ελλάδα, στα, στους καταβλισμούς. Τα χειρότερα πράγματα έχουν γίνει και έχουν συμβεί στις οικογένειές τους. Δεν έχουν καμία ψυχολογική υποστήριξη. Τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν. θα είναι ισορροπημένοι ενήλικες, αλλά να τις βοηθήσουμε γρήγορα. Να μην αναφέρω καν την κατάσταση των κοριτσιών που έχουν υποστεί βιασμούς. Και τι γίνεται στα hot spots. Τι γίνεται με τα παιδιά εκεί. Στη Λιβύη, για παράδειγμα. Πρόσφατα με ενημέρωσαν ότι στα πλαίσια προγράμματος του ΟΗΕ, ένα μεγάλο αριθμό ε, παιδιών από τον Παγκλαντές, από τον Ναϊρόμπι. Αυξάνεται. Λαμβάνεται αυτό υπόψη. Και φυσικά η πλέον δραματική κατάσταση για μένα είναι η κατάσταση των νεαρών Αφγανών, τους οποίους τους αντιμετωπίζουν ως μετανάστες και πάλι πέφτουν θύματα τη χείρη τη κατάχρηση. Γιατί δεν μοιάζεται κανεί να του βοηθήσει. Και φυσικά ξέρουν ότι πρέπει να αποφύγουν ε, την καταχώρηση και προφανώς είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι οποιοδήποτε άλλος να καταστούν εργαλεία εγκληματικών και τρομοκρατικών οργανώσεων. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Άννα, να κάνω μια πρόταση στην Κιάρα και στον Στίβεν από τις δύο γενικές διευθύνσεις. Την επόμενη φορά θα οργανώσουμε τη συζήτηση αυτή σε πιο ευνοϊκή χρονική θηρίδα για να έχουμε πιο πολλοί συναδέλφους μαζί μας. Γιατί το θέμα αυτό άπτεται και πολλών άλλων ζητημάτων και προφανώς θα είναι πολύ ενδιαφέρον να τα συζητήσουμε όλα αυτά και διαπιστώνουμε πόσο προβάλλεται στον τύπο, στη δημοσιότητα το θέμα αυτό. Η περιπλοκότητα ωστόσο του ζητήματος είναι μεγάλη. Το σύστημα ασύλου, το σύστημα κράτησης, υπάρχουν και πραγματικά κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα ενοποίησης τα οποία περιλαμβάνονται. Ας φροντίσουμε λοιπόν να είναι πιο ευνοϊκή η χρονική στιγμή την επόμενη φορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Κόμες και την κυρία Κινίτσι, οι οποίοι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν προφανώς το θέμα αυτό. Γιατί χρειαζόμαστε μεγάλη πολιτική υποστήριξη. Θα συνεχίσουν να το παρακολουθούν λοιπόν και να είναι σε επαφή μαζί μας για την επόμενη χρονική στιγμή που θα διοργανωθεί συζήτηση με πιο πολύ συμμετοχή. Δεν έχει νόημα να ξεκινήσει μια καινούργια συζήτηση στην παρούσα φάση. με μόνο εμένα και την Άννα ως βουλευτές. Παρά το γεγονός ότι φυσικά θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να παρακολουθούμε το πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Σας ευχαριστούμε για την εξαιρετική παρουσίαση, για τη δουλειά σας και σας ευχόμαι καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στις μελλοντικές σας εργασίες. Σας ευχαριστούμε και σας Άννα. Ευχαριστούμε λοιπόν και όλους τους υπαλλήλους και όλους τους υπόλοιπους. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. That's the end of the meetings. Και έτσι ολοκληρώνεται η συνεδρίαση. Πέρας. Επόμενη συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου στο Στρασβούργο.